Meine sehr verehrten Damen und Herren. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας καλωσορίσω και χαίρομαι ιδιαίτερος διότι ε, μπορώ να σας υποδεχτώ εις την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών σε μία ακρόαση και ο συνάδελφος Λούκας Αγγιλάρα ήρθε εξαιρετικά εδώ διότι αυτό το θέμα νομίζω ενδιαφέρει πλέον όλους διότι πριν από λίγα χρόνια κοιτούσαμε με έκπληξη τα πιο περίπλοκα, τους πιο περίπλοκους υπολογιστές νέας γενιάς βλέπουμε τώρα ότι η τεχνολογία ναι μεν συνεπιφέρει πολλές δυνατότητες αλλά και πολλούς κινδύνους ε, για να δραστηριοποιηθούν εγκληματίες Δηλαδή, πού πρέπει κανείς να τραβάει τη γραμμή, ποιες είναι οι ε, προϋποθέσεις. Είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα και θα ακούσουμε μία σειρά από εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας δώσουν ε, μία καλύτερη εικόνα για το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις και πώς μπορεί ε, να ακολουθήσει νέες προτάσεις. Βέβαια ε, για αυτό υπήρξε έναυσμα το σχέδιο και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία οδηγία σχετικά με ε, τους ε, υπολογιστές και αυτό έχει ε, οδηγήσει σε συζητήσεις και σε άλλες επιτροπές, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και άλλες και γι' αυτό χαίρομαι ότι είναι εδώ η συνάδελφος Κριστίνα Όγιουλαντ από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και συγχρόνως η συντάκτρια, ο συντάκτης μάλλον Κρίσια από την Επιτροπή Ήτρε και εφόσον αυτή η πρόταση της Επιτροπής για μια, οδηγία, για μια οδηγία δημοσιεύτηκε πέρυσι το φθινόπωρο κάθεται δίπλα μας και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον οποίο είχαμε έκτοτε συζητήσεις και έτσι θα αντικατασταθεί η οδηγία που είχε ψηφιστεί στο Συμβούλιο το 2005 και ε, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συζήτηση. Όταν κοιτάτε λοιπόν προς τα έξω βλέπετε ότι υπάρχει ο κύριος Μίλλερ από το Υπουργείο Εσωτερικών υπεύθυνο για την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά καθημερινά για να κάνω μία σύντομη εισαγωγή. Από την αρχή του χρόνου συζητάμε το θέμα αυτό και ήδη υπάρχουν ορισμένες συζητήσεις μεταξύ ε, διαφόρων ε, μελών επιτροπών. Το ε, Συμβούλιο παρουσίασε τη θέση του τον Ιούλιο και έκτοτε προέκυψαν ορισμένα προβλήματα, δηλαδή αν ε, οι, κυβερ... οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι ε, ο βασικός λόγος για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σε αυτό το χώρο. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στι οδηγίες μας και τι θα γίνει με τα θέματα τις οποίες ε, δεν έχουμε ακόμη αντιμετωπίσει, δηλαδή το cloud πλούτη να ε, είναι κανείς στο διαδίκτυο και ε, να ε, πετάει συγχρόνως σε ένα αεροπορικό ταξίδι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να μεταδοθούν και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες που ανταποκρίθηκαν ή στην πρότασή μας διότι έτσι θα έχουμε μία επικοδομητική συζήτηση. Η δομή μας θα είναι ως εξής. Το πρώτο μέρος ε, θα ε, προεδρεύσει η Κριστίνα Όγιουλαντ ε, για το ποιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης, σε ποιο επίπεδο κρατών μελών και σε ποιες σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα και με ποιον τρόπο μπορούν να προλαμβάνονται οι κυβερνοϋποθέσεις. Το τρίτο είναι η συνεργασία και το τέταρτο η προστασία των δεδομένων και νομική ασφάλεια. Υπάρχουν βέβαια διάφορες δυνατότητες αλλά θα παρακαλούσα εάν ε, υπάρχουν ερωτήσεις να ε, έχουμε ερωτήσεις σύντομες και όχι μεγάλες δηλώσεις διότι θέλουμε να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Αν θέλουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας μπορούμε να το κάνουμε ανα πάσα στιγμή και θα έχουμε ακόμη πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για αυτή την εργασία αλλά τώρα πρέπει ιδίω να δώσουμε τον λόγο στους εμπειρογνώμονες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ενδεχομένως θέλουμε να τους κάνουμε. Θα υπάρχει 10 λεπτά για τους ομιλητές και ένα λεπτό για κάθε ερώτηση. Και δίνω το λόγο στην Κριστίνα Όγιουλαντ για να προεδρεύσει για το πρώτο μέρος. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι και προσκεκλημένοι. Ήρθαμε, μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να συζητήσουμε το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων και από την κάθε χώρα αλλά και στο σύνολο. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που προεδρεύω σε αυτό το πρώτο γύρο των συζητήσεων διότι και εγώ είμαι από την Εσθονία και γνωρίζετε όλοι καλά ότι το 2007 η Εσθονία βίωσε μία τεράστια κυβερνοεπίθεση. Μερικοί μίλησαν και για κυβερνοπόλεμο και γι' αυτό έχουμε εμπειρίες που θέλουμε να μοιραστούμε με άλλες χώρες. Προσωπικά εγώ ενδιαφέρομαι να σας ακούσω τις απόψεις σας ως εμπειρογνώμονες σήμερα στην ακρόασή μας. Είμαι πεπισμένη ότι πολλοί και πολλά όργανα συμφωνούν ότι χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία για να αντιμετωπιστεί το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων και μάλιστα εναρμόνιση της νομοθεσίας και των δραστηριοτήτων μας για να προστατεύσουμε τις στρατηγικές μας υποδομές καθώς και την, να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Τέλος, για την σύντομη αυτή εισήγηση θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο τα στενά όρια του τίτλου που, προτείναμε, αλλά και ευρύτερα για τις πολύ ευρύτερα πώς να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα αυτό και μέσα και έξω από τα σύνορα της Ένωσης. Τι δραστηριότητα πρέπει να αναλάβει η Ένωση και μέσα της και διεθνώς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσέλευσή σας και ξαναδίνω την Προεδρία και το λόγο σε σας Και εμείς στον Ιάκουμ Μπορατίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που καλέσατε την Κομισιόν σε αυτή την ακρόαση γνωμόνων, Η κυρία Λέντ ε, μας, ε, ε, οδήγησε στο να αναλάβει η Κομισιόν αυτή την πρωτοβουλία για να παρουσιάσει μια πρόταση νέας οδηγίας για τις επιθέσεις ε, κατά των συστημάτων πληροφορικής, ε, οι επιθέσεις κατά της Εστονίας μας εκανε να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να δώσουμε μια απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό η νέα πρόταση και θα επικεντρωθώ σε αυτή γιατί θα αναφερθούμε στις απαντήσεις που δίνονται κατά του εγκλήματος στον κυβέρνο χώρο. Υπάρχει λοιπόν μία ολόν και μεγαλύτερη απειλή από τις κυβερνοεπιθέσεις ε, πιο πρόσφατα. Η Α.Ι.Οκτά της ε, Europol έχει βεβαιώσει ότι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος ε, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ίντερνετ και τα λεγόμενα botnet, τα δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ, για να διαπράξουν και άλλα είδη κυβερνοεγκλημάτων. Ο συνολικός στόχος της υγείας είναι ε, να μειώσει τον αριθμό ε, και τη συχνότητα των επιθέσεων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός ε, και στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένο στόχος είναι να καταδικαστούν οι εγκληματίες μέσω της προσέγγισης του ποινικού δικαίου να βελτιωθεί η διασυνεργειακή συνεργασία μεταξύ των βιωτικών αρχών και να υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης αποτελεσματικά και συλλογής δεδομένων. Αυτό σχετίζεται πιο συγκεκριμένα στο να αυξηθεί το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι πολύ μικρό. Επίσης εισάγονται νέες επιβαρυντικές περιστάσεις. Καταρχήν, η πράξη χρησιμοποίησης botnet ή παρόμοιου εργαλείου ε, βοήθησε την οργάνωση επιθέσεων μεγάλης ε, κλίμακας ε, και αυτό είναι επιβαρυντική περίσταση και δεύτερον έχουμε και τις λεγόμενες spoofing attacks ε, όπου οι δράστες κλέβουν την ταυτότητα κάποιου άλλου και τα χρησιμοποιούν και ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η πρόσφατη πρακτική να στέλνει κάποιο email ε, με προσαρτήματα που, ε, φαίνεται ότι προέρχονται από κάποιον ε, άλλον και δυστυχώς και στην Κομισιόν παρά την προστασία του μηχανισμού προστασίας που έχουμε και τα διάφορα φίλτρα περνάνε τέτοιου είδους email. Επίσης, στην πρόταση αυτή έχουμε εισαγάγει μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη για να απαντήσουν σε έκτακτο αίτημα από το δημοσίο και τον ιδιωτικό τομέα μέσω του δικτύου επαφών 24 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις. Και τέλος, ε, καθώς έχουμε άγνοια σε σχέση με την κλίμακα, με το μέγεθος του προβλήματος, και τις συγκεκριμένες περιπτώσει, όπου λαμβάνουν χώρα τέτοιες επιθέσεις ε, υπάρχει μια πρόβλεψη να υπάρχει ένας μηχανισμός να συλλέγουν δεδομένα τα κράτη-μέλη για τις κυβερνοεπιθέσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πλήρως ότι δεν πρόκειται αυτή αυτή η νομοθεσία δεν απαντά πλήρω ε, στο πρόβλημα. Πρόκειται απλώ για ένα νομοθέτημα σε μια σειρά λοιπόν νομοθετημάτων που μπορούν να μα βοηθήσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσουμε καλύτερα συλλογικά στι απειλέ που προκύπτουν από το κυβερνό έγκλημα. Να υπενθυμίσω ότι η στρατηγική εσωτερική ασφάλεια στη σχετική ανακοίνωση τη Κομισιόν που υιοθετήθηκε Νοέμβριο που κατέστησε την καταπολέμηση του εγκλήματος ένα από τους κύριους στόχους και πιο συγκεκριμένα μέτρα όπως τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ε, κέντρο κατάρτισης καθώς ε, και εταιρική σχέση δημοσιοδιωτικού τομέα. Αυτά αναφέρονται ως κύρια μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση και θα έλεγα ότι το σημερινό εγχείρημα που ελπίζουμε να βοηθήσει στη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του κλίματος στον κυβερνό χώρο είναι ένας τρόπος να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τίθεται από αυτή τη συνεδρία, δηλαδή ποιο είναι το σωστό επίπεδο απάντησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατημέλη κτλ. Η Κομισιόν ε, τώρα υλοποιεί μια μελέτη σκοπιμότητας και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε μια σειρά ερωτήσεων που θα πρέπει να βρίσκεται αυτό το κέντρο, ποια θα πρέπει να, ποιες θα πρέπει να είναι οι λειτουργίες του, πώς θα σχετίζεται ε, με τις ικανότητες σε επίπεδο κρατών μελών και πώς συνολικά μπορεί να απαντήσει καλύτερα στις ανάγκες. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία μέσω της οποίας ε, προσπαθούμε να βρούμε μια λεπτομερή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Επίσης, να αναφέρω κάποια άλλα θέματα που ενδεχομένως να αναφέρουν και κάποιοι άλλοι ομιλητές. Ένα θέμα για μας, για την γάμα δελτα ιστορικών υποθέσεων, είναι πώς θα προωθήσουμε την ικανότητα εφαρμογής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τέσσερα χρόνια η Κομισιόν προσπαθεί να αναπτύξει καινοτόμε προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την κατάρτιση για την κατηπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να γεφυρώσουμε τους διάφορους κόσμους αφενός ε, ιδιωτικών αρχών και αφετέρου δημοσίου ε, συγγνώμη, ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των ΣΕΡΤΣ, ε, αυτών των ε, ομάδων ε, που απάντηση απάντησης σε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Αυτά για να δώσουμε αποτελεσματική απάντηση στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Και φυσικά κάτι άλλο που διερευνούμε είναι το θέμα της διεπαφής του κέντρου Τώρα, διακυβέρνηση του διαδικτύου, τεράστιο θέμα, το οποίο υπερβαίνει τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε σωστά προκειμένου να εξισορροπήσουμε μεταξύ της διασφάλειας, υπάρχει ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της ελευθερίας και της ασφάλειας και εμπιστοσύνη. Ένα θέμα που έχουμε στην ημερική διαταξή μα είναι η πρόθεση των συστάσεων επιβολή τη νομοθεσία ό,τι αφορά την πρόληψη τη κατάχρηση των κριτικών υποδομών του διαδικτύου. Οι συστάσει έχουν υποστηριχθεί διεθνώ στο ΙΚΑΝ από τι κυβερνήσει ε, και αυτό είναι ένα θέμα που βρίσκεται και στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων ομάδων που εργάζονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό για μας είναι διάφορα μέτρα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο ίντερνετ. Είμαστε στο τελικό στάδιο θέτησης της για το θέμα αυτό. Έχουμε μεγάλο βαθμό συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και έχουμε και το πρόγραμμα το πιο, πιο ασφαλές διαδίκτυο που τρέχει υπό τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Information Society, κοινωνία των πληροφοριών, όμως ε, όλα αυτά ανήκουν σε μια συνολική απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε για την καταπολέμηση του κλίματος στον χώρο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, ενώ συζητούμε το μέλλον αυτής της οδηγίας, κατά κάποιο τρόπο να μην ε, προσπαθήσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του ποινικού δικαίου να βρούμε μια πανάκια σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Προφανώς εδώ δίνουμε μια συγκεκριμένη απάντηση μέσω του δικαίου. Αλλά φυσικά θέλουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για πολλά άλλα μέτρα που δεν είναι και νομοθετικού χαρακτήρα. Αλλά είναι καθοριστικά για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο κυβερνό έγκλημα. Ελπίζω να μην ξεπεράσει και το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μποροτσίνσκι για αυτή την εισαγωγή σας. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι με την πλευρά της, στην πλευρά της Κομισιόν γιατί αναγνωρίζει και αυτό την ανάγκη να διευθετηθεί ο κυβερνοχώρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή μας που εκπροσωπεί την Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας αυτή την ακρόαση. θα σας παρουσιάσω την άποψη του Συμβουλίου. Πράγμα που μου διευκόλυνε πολύ ο συνάδελφος της Κομισιόν που ήδη παρουσίασε μια σειρά μέτρων που προτείνονται. Όλοι συμφωνούν, δεν χρειαζόταν ακρόαση γι' αυτό, ότι η απειλή αυξάνεται. Είναι διαμεθοριακή και πρέπει να απαντηθεί πανενοσιακώς. θα ήθελα να τονίσω ότι το Συμβούλιο προετοιμάζει με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν μία σφαιρική ανταπόκριση. Υπάρχει το ψηφιακό πρόγραμμα για την Ευρώπη, το πρόγραμμα δράσης για την ασφάλεια στο ίντερνετ και ολόκληρη σειρά μέτρων που συζητιούνται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και θέματα όπως η δημιουργία ενός κέντρου για την αντιμετώπιση των κυβερνοεγκλημάτων και αναμένουμε να προταθούν τον Οκτώβριο προσαρμογές της ισχύουσας αυτής νομοθεσίας. το επόμενο βήμα θα είναι θα υποβληθεί φέτος. Είμαστε πεπισμένοι ότι αφόσον εφαρμοστούν τέτοιου είδους μέτρα θα βελτιωθεί η ανταπόκριση, η δυνατότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει το κυβερνοέγκλημα. Η οδηγία για την καταπολέμηση των επιθέσεων έναντι πληροφοριακών συστημάτων είναι τμήμα της όλης αυτής στρατηγικής και νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο βήμα της απάντησης, της ανταπόκρισης μας αφορά το θέμα του ορισμού των εγκλημάτων ή παραπτωμάτων, τις κυρώσεις, τις επιβαρυντικές συνθήκες και ολόκληρη σειρά ποινικών μέτρων που θα είναι η απάντησή μας προς τα εγκλήματα αυτά. Βασίζεται στο άρθρο 83 της συνθήκης ε, και έχει σαφή στόχο και εύρος. Γνωρίζετε και έχει υποθεί και προηγουμένως ότι το Συμβούλιο έκανε πολύ έντονες συζητήσεις υπό την Ουγγρική ήδη Προεδρία. Σήμερα, αν δεν απατώμε, είναι ακριβώς ένας χρόνος μετά την πρώτη ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλειών και τον Ιούνιο του 2011 είχε ήδη επιτευχθεί μία σύγκληση θέσεων των χωρών μελών να σας πω ποιες είναι οι κύριες αρχές της εξέτασης αυτού του σχεδίου οδηγίας. Τέσσερις κύριοι άξονες. Ο πρώτος να παραμείνει βασικά η πρόταση της Κομισιόν και να συμπεριλάβει και, και επιθέσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Χρειάστηκε να λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορές των νομικών και δικαστικών συστημάτων των χωρών μελών δεύτερων. Εξισορρόπηση μεταξύ κυρώσεων προσπαθήσαμε να απορρίψουμε ελάσσονα παραπτώματα και να περιοριστούμε σε τα πιο σοβαρά. Τρίτον, προσπαθήσαμε τη γλώσσα της οδηγίας να την κρατήσουμε όσο το δυνατόν ουδέτερη, πιο ουδέτερη και τεχνική γινόταν. Διότι οι απειλές που αποτελούν αυτές οι ε, επιθέσεις αυξάνονται και η γενικότερη ιδέα είναι όπως είπα να παραμείνει τεχνικό και ουδέτερο το κείμενο. Τέλος, να παραμείνουμε συνεπείς με πρότυπα που έθεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στη λεγόμενη συνθήκη της Βουδαπέστης. Ελπίζω να συμμερίζεστε τις αρχές και τους στόχους αυτούς και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για την εξέταση του σχεδίου οδηγίας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. γιατί την επεξηγηματική έκθεση εν ονόματι της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζάστιν Μίλε σχετικά με την, ε, ε, τον προϊστάμενο πολιτικής για την αντιμετώπιση εγκλήματος στον κυβερνοχώρο από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και με συγχωρείτε δύο λεφτά μέχρι ότου ευθυγραμμίσω την τεχνολογία. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να ευχαριστήσω την κυρία Χολμάγερ που οργάνωσε αυτή την ακρόαση γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας και ιδίως την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να σας πω το τι βλέπουμε και ε, πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε διορθωτική δράση διότι πρέπει να σας πω ε, τι <clears throat> πώς αντιμετωπίζει το κυβερνοέγκλημα το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα και η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 650 εκατομμύρια ε, λίρες για τέσσερα χρόνια για να προστατεύσει τον κυβερνοχώρο από το έγκλημα και να μπορέσει να έχει τις αναγκαίες ε, σωστές δράσεις. Ε, όλοι είμαστε υπεύθυνοι να επιλύσουμε τα προβλήματα που, βρίσκουμε, που αντιμετωπίζουμε στον κυβερνοχώρο διότι όλοι εποφελούμαστε είτε είναι για τον ιδιωτικό τομέα είτε για το, τις κυβερνήσεις όλοι εποφελούμαστε. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχουν διάφορες ε, ε, τάξεις της κοινωνίας που θα πρέπει να συμβάλλουν στο να έχουμε έναν πιο ασφαλή κυβερνοχώρο. Χρειάζεται λοιπόν και μία διεθνής ευθύνη. Ε, διότι πρόκειται για διεθνή εγκληματικότητα και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε σε όλους τους τομείς, στον τομέα της κοινωνίας, στον τομέα της ε, εφαρμογής της ε, νομοθεσίας για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Τι θεωρούμε ότι είναι οι βασικές εθνικές ευθύνες. Καταρχήν, κάθε κράτος πρέπει να έχει τις σωστές ε, νομοθετικές αντιδράσεις, δηλαδή να μπορεί να ε, πατάξει το κυβερνοέγκλημα ε, έχοντας συγκεκριμένες επιθετικές μεθόδους. Μιλήσαμε πολύ για την οδηγία και πόσο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και στηρίζουμε την κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά δεν αναφερόμαστε μόνο στην εθνική νομοθεσία αλλά και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς σε εθνικό επίπεδο την νομοθεσία να την χρησιμοποιήσουν τα, οι, οι αστυνομικές δυνάμεις και ε, επίσης είναι ένα είδος εργασίας το, οποίο πρέπει να βελτιωθούμε και στην επόμενη τετραετία στο Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο θα δημιουργήσουμε ειδικέ μονάδες αλλά να, θα μεταδώσουμε την γνώση του τι είναι το κυβερνοέγκλημα και πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων δυνάμεων διεθνώς πατάξεως του, του κυβερνοεγκλήματος. Πρέπει λοιπόν πρώτον να ξέρουμε τι είναι το πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς μπορεί οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας και το κοινό να συνεργαστούν για να προστατευθούν όλοι. Έχουμε μία προσέγγιση ε, για συνεργασία. Δεν μπορεί κάθε τομέας να προχωρήσει μόνος του, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και όταν ε, αυτό το, εφαρμόσουμε σε διεθνές επίπεδο αντιλαμβανόμαστε ότι στα πλαίσια της ε, συνθήκης της Βουδαπέστης πρέπει να υπάρχει διεθνή συνεργασία προς τους στόχους τους οποίους έχουμε ήδη καθορίσει. Χαιρετίζουμε την εργασία η οποία γίνεται στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, δεν συμμετείχαμε ε, στη συζήτηση αυτής της οδηγίας και είπαμε ε, σαν Ηνωμένο Βασίλειο το πρόβλημα είναι διεθνές και στηρίξαμε το κείμενο της οδηγίας που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο του Ιουνίου θεωρούμε ότι ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ένας ρόλος συντονιστικός και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιαστεί εις ε, την αντίδραση των δυνάμεων αφαρμογής ε, του νόμου και ε, να υπάρξει συνδυασμός με ε, άλλα μέτρα όπως η συνεργασία μεταξύ δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα ε, με συνεργασία με διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η ICAN για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα του κυβερνοχώρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά και με τις Ηνωμένε Πολιτείες και το χαιρετίζουμε αυτό και επιπλέον ε, πρέπει να υπάρξει μία προώθηση σε όλα τα κράτη-μέλη ε, του θέματος αυτού. Για να συνοψίσω λοιπόν. Όπως σας είπα, στηρίζουμε την ε, διεθνή συνεργασία για να επιλύσουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Θα συνεργαστούμε με άλλα κράτη-μέλη και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με άλλες χώρες για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό ε, και ε, θα μεταδώσουμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας προς άλλες χώρες ε, διότι εφόσον θα ξεκινήσει το πρόγραμμα τον Νοέμβριο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τη βάση συνεργασίες με πολλές κυβερνήσεις, με πολλά κλιμάκια της κοινωνίας για να μπορέσουμε ε, να επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να σας παρουσίασα τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μίλλερ για την έκφραση της άποψής σας. Τώρα η κυρία Χέιλι Ντιέρ Μακλόρ που είναι και αυτή η Εσθονή και έχει συνεργαστεί με τα όργανα του ΝΑΤΟΥ Καλό σας απόγευμα. Θα σας παρουσιάσω την ε, άποψη της ιστονικής κυβέρνηση για την ε, ασφαλεία στον κυβερνοχώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες επιθέσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τι συνέβη το 2007 και τι συνέβη από το 2007 και μετά στην Ευρώπη. Το 2007 βιώσαμε ε, τέτοιες επιθέσεις ε, πολιτικού χαρακτήρα, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε μεγάλο βαθμό και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε μόνοι μας. Δεν υπήρχε διεθνής μηχανισμός για να μας βοηθήσει. Οι, κάποιοι επαγγελματίε ε, τεχνολογίες των πληροφοριών ήξεραν άλλους άλλες χώρες και μας βοήθησαν ε, για να υπάρχει διεθνής αρρωγή στην Εστονία κατά το 2007 για να αντιμετωπιστούν και βρουν επιθέσει, Έτσι λοιπόν ε, ήταν επιτυχής αυτή η διαδικασία. Έτσι λοιπόν προετοιμαστήκαμε σε χώριο επίπεδο και μπορέσαμε να ενεργοποιήσουμε τη διεθνή υποστήριξη κατά τον, ε, τη διάρκεια των τριών αυτών εβδομάδων. Και ποια είναι τα διδάγματα από τις επιθέσεις του 2007. Καταρχήν ότι κάποια, κάθε χώρα θα πρέπει να έχει συστήματα προστασίας ε, των ΣΔΙΤ ε, και αυτό είναι ο ακραγωνίας λήθος ε, της ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Επίσης, μηχανισμοί διαχείρισης ε, κρίσεων ε, και θα, θα πρέπει να υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν και διάφορα νομοθετήματα. Και το δεύτερο δίδαγμα ήταν ε, ότι η διεθνή συνεργασία και συντονισμός είναι βασικά αν θέλουμε να... αν πρόκειται να βιώσουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Από το 2007 υπήρξαν πολλές εξελίξεις στο διεθνή τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί πολλές πρωτοβουλίες. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια ευρία προοπτική σε σχέση με το τι κάνουν οι υπόλοιπε διεθνείς οργανισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ποιο είναι ο συγκεκριμένο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είδαμε από τότε να ξεφυτρώνουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και οι διεθνείς οργανισμοί μέχρι τώρα φαίνεται να βρήκαν το ρόλο τους ε, και την διαγορά τους σε αυτό το τεράστιο τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Δεν θα ξεκινήσω με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εσείς μάλλον θα γνωρίζετε τις περισσότερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα ξεκινήσω σε παιδό ΙΕ. Είχαμε μία έντονη συζήτηση στην Επιτροπή Εφοπλισμού στα Ηνωμένα Έθνη, όπου πέρασαν ε, κάποια ψηφίσματα σε σχέση με το να χρησιμοποιείται η ασφάλεια των πληροφοριών ε, ως ε, κακόβουλα εργαλεία κατά άλλων χωρών. Έτσι λοιπόν το 2010 η ομάδα εμπειρογνωμόνων στον ΟΗΕ ε, πόνισε μια έκθεση που έλυσε πολλά θέματα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και τώρα μπορούμε να πούμε Είπαμε ότι η διεθνή νομοθεσία που διέπει την ε, διεθνή χρήση αυτής ε, της σε έναντι άλλων χωρών ισχύει και για τον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν ε, ο νόμος, η νομοθεσία των ένοπλων σειράξεων ισχύουν και για τον κυβερνοχώρο. Δηλαδή υποτίθεται ότι οι χώρες δεν μπορούν να επιτεθούν στον πληθυσμό, μη στρατιωτικό πληθυσμό ή σε μη στρατιωτικές υποδομές και στον χώρο και τα δευτερογενή και τριτογενή αποτελέσματα ε, είναι ότι θα πρέπει να απόσχουν αυτές οι χώρες από το να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία στον κυβερνοχώρο. Κάποιες ε, χώρες ε, δικτατορικές θα ήθελαν να έχουν να επιδίδονται σε πόλεμο στον κυβερνοχώρο, ε, κάτι που δεν το επιθυμούμε και ε, θα ήθελαν κάποιες συνθήκες ε, για να μπορούν να ασκούν περισσότερο έλεγχο στον πληθυσμό τους και φυσικά οι δυτικές δημοκρατικές, τα δυτικά δημοκρατικά καθεστώτα δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και εδώ περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένα άλλο συμπερισμό πολύ σημαντικό από την έκθεση του είναι ότι η αυτοάμυνα των χωρών επιτρέπεται στον κυβερνό χώρο σύμφωνα με τη χάρτα του ΟΗΕ. Τώρα, προχωρώ. Το ΝΑΤΟ έχει υιοθετήσει δύο πολιτικές για την προστασία των στρατιωτικών υποδομών και των υποδομών του ΝΑΤΟ στις διάφορες ε, χώρες. Δεν προβλέπει το ΝΑΤΟ υποδομές, ε, μάλλον προστασία των ε, μη στρατιωτικών υποδομών. Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ εστιάστηκε σε πιο αντιδραστικά μέτρα, αν κάτι συμβεί, θα μπορέσει το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει τη συλλογική άμυνα, αλλά αυτό είναι ε, αντικειμένο πολιτικής απόφασης. Δηλαδή, αν ε, υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις ε, κατά του ΝΑΤΟ, τότε θα θεωρηθούν ένοπλες επιθέσεις. Θα ισοδυναμούν με ένοπλες επιθέσεις, αλλά το ΝΑΤΟ δεν λέει πότε μπορεί να ληφθεί αυτή η πολιτική απόφαση και αν ε, έχουμε μια ευρύτερη σύραξη και κυβερνοεπιθέσεις, τότε θα υπάρχει απάντηση και μπορεί να υπάρχει και μια απάντηση συλλογικής άμυνας. Αυτό ήταν το κύριο αποτέλεσμα της πολιτικής που θετήθηκε τον ε, Ιούνιο, κατόπιν έχουμε τον ε, ΟΣΑ, ΟΣΑ, είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπόρεσε να δώσει στην κοινότητα την προσέγγιση soft law. Ο ΑΣΕ, με συγχωρείτε, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, στον κυβερνοχώρο χρειάζονται για να παρεμποδίσουμε ε, κάποια παρεξήγηση των προθέσεων των χωρών. Έτσι λοιπόν θα υπάρχουν μέτρα διαφάνειας, ε, σημεία επαφής και όλα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν σε δύο-τρία χρόνια και ο ΑΣΕ άρχισε την αναπτυξή τους. Στη συνέχεια έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Μέχρι τώρα είναι το πιο σημαντικό νομοθετήμα στον τομέα αυτό γιατί σκοπεύει να εναρμονίσει το νομικό συστήματα των συμμετέχοντων χωρών, συμμετέχοντων χωρών και διαθέτει όλες τις κυρίες αρχές για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Δεν χρειαζόμαστε ουσιαστικά άλλε διεθνείς συμφωνίες. Αν όσοι χώρες στον κόσμο διαθετούσαν τις αρχές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, τότε θα ήμασταν καλυμμένοι. Και εδώ μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατόπιν έχουμε τον ΩΣΑ, ο οποίος έχει... Ε, Μία σκουπιά έχει μάλλον κάποιες υποδομές περισσότερο οικονομικού χαρακτήρα και έχει κάποιες ε, συστάσεις αλλά στα χαρτιά. Έτσι λοιπόν, ε, σε όλες αυτές τις διεθνείς πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον κατάλληλος οργανισμός για να επιλύσει όλα τα θέματα του εγκλήματος του κυβερνοχώρου στα δικά της μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον πυλώνα της κοινή ασφάλειας και άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή νομοθεσία και έχει αρμοδιότητες δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Επίσης έχει νομοθεσία για την εσωτερική αγορά. Κανένας άλλος οργανισμός στον κόσμο δεν έχει τέτοια εντολή για να αντιμετωπίσει θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν, μάλλον θα, θα ακούσουμε περισσότερα σήμερα για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χαίρομαι ήδη που το 2009 η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Information Society ξεκίνησε μια πολιτική για την προστασία ε, των κριτικών υποδομών ε, και τώρα έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών ε, και ετοιμότητα. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ιστορικών Υποθέσεων πρότεινε ένα καλό νομοθέτημα που το συζητούμε εδώ σήμερα και αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος και υπάρχουν και πολλές άλλες καλές πρωτοβουλίε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει αλλά τι μας λείπει πιθανότατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συνολική εικόνα γιατί θα πρέπει να γίνει στην ασφαλεία στον χώρο και ο συντονισμός μεταξύ αυτών των διάφορων πρωτοβουλειών, οι οποίες είναι όλες πολύ καλές. Λοιπόν, για να φτάσω τώρα στη σημερινή νομοθεσία και στο σχέδιο κειμένου, αυτό είναι ένα μεγάλο κύμα, βήμα προς τα μπρος, εναρμόνιση της απάντησης των κρατών μελών και εναρμόνιση των ε, κυρώσεων, των ποινών, είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά ε, είναι αποτρεπτικό εργαλείο. Κάποιες από αυτές τις ε, οργανώσεις που προβαίνουν σε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο είναι πολύ πιο ισχυρέ από τι εθνικέ αστυνομίε. Πρέπει λοιπόν να γίνει πολλή δουλειά και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενδυναμωθεί και η διεθνή και η εθνική αλλά ε, και η διεθνή διάσταση του συντονισμού και της συνεργασίας. Ε, αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προβλέψει κάποιο σύστημα επαλήθευσης ότι αυτές οι ιδέες που ακούτε εδώ θα εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τώρα τις ΔΙΤ, τις ε, συμπράξεις τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες συμπράξεις, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν κάτι παρόμοιο και νομίζω ότι εμεί στην Ευρώπη πρέπει να τις αντιγράψουμε. Οι μεγάλε εταιρείε στην Ευρώπη δέχονται καθημερινά επιθέσει. και λόγω αυτών των επιθέσεων έχουν οικονομικέ απώλειε και πιθανότητα θα έχουν τι καλύτερε πληροφορίε ε, για το τι συμβαίνει και έξω και ποιο του επιτίθεται, ποιοι είναι οι δράστε. Και ο ιδιωτικό τομέα έχει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει σήμερα σε οποιαδήποτε απάντηση για την καταπολέμηση του κυβερνών κλίματο. Επίση, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Πολύ σημαντικό αν ε, ο μηχανισμός αυτός ε, τεθεί σε λειτουργία, τότε θα είναι πολύ πιο ασφαλής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερα και τι κάνει ε, τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τώρα δεν έχουμε την νομοθεσία CAP σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάποια τμήματα εδώ και εκεί, αλλά δεν ξέρω πόσο τελεσματικά έχουν συμπεριληφθεί στην συνολική εικόνα, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό σήμερα. Στα εξωτερικό προσκήνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες που δεν έχουν τα μέσα, ίσως ε, και με οικονομικά, αλλά και με άλλα μέσα, γιατί τελικά είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση και δεν υπάρχουν σύνορα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν, πολλέ από τι απειλέ προέρχονται, πηγάζουν από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όμορε χώρε και θα πρέπει οι οικονομίε να σκεφτούν ε, τι θα κάνουν με τι λιγότερο προηγουμένε χώρε που είναι γύρω μα ή αλλού για να τις βοηθήσουν ε, να οικοδομήσουν ε, την ικανότητα τους γιατί τελικά αν αφήσουμε αυτούς τους παραδείσους να αρθίσουν στον κόσμο τελικά θα μα επιτεθούν και εμά. θα μπορούσε και άλλα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πώ θα μπορούσε να προστατεύσει και τι δικέ τη πληροφορίε και τα δικά τη όργανα, του δικού τη θεσμού. αλλά γενικά θεωρώ ότι οδεύουμε στη σωστή κατεύθυνση και εκ μέρους της κυβέρνησης της Εστονίας χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ασφαλή στον κυβερνοχώρο έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ε, πλήρη επισκόπηση του τι κάνουν οι διεθνείς ε, οργανώσεις και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας διότι είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Τώρα ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κύριος Μιχάλ Ζαλεύσκη ο οποίος Α, μετακινηθήκατε βλέπω. Ε, θα αναφερθεί εις ε, τις ε, εμπειρίες της πολωνικής αστυνομίας. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. εκπρόσωπο. την μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της πολωνικής αστυνομίας και θα ήθελα να σας δείξω πώς είναι τα πράγματα στην Μπολονία. Οι πρώτες δομές ε, για την καταπολέμηση αυτή στην εθνική αστυνομία δημιουργήθηκαν το 1996. Έχουν αυξηθεί δυναμικά οι αριθμοί των επιθέσεων αυτών και Γι' αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί τέτοιου είδου μονάδες μέσα στα πλαίσια της αστυνομία και αλλού. Πριν από ένα χρόνο, την 1η Ιουνίου του 2010, δημιουργήθηκε η υπομονάδα στην οποία εργάζομαι. Είναι, βρίσκεται στο κτίριο, στο κεντρικό κτίριο της αστυνομίας και εδώ βλέπετε τη δομή της μονάδας μας. Έχουμε 26 αστυνομικούς εκεί. Ιδού τα κύρια καθήκοντα της μονάδας ταυτίζει και παρακολουθεί τους τομείς του κυβερνοεγκλήματος συνεργάζεται με διοικητικούς και με ιδιοκτήτες ε, δικτύων, ηλεκτρονικών δικτύων και είμαστε υπεύθυνοι για την ταύτιση και την επιβολή του νόμου κατά των εγκληματιών που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε νέα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε το κυβερνοέγκουλημα. ή να βελτιώσουμε τη συνεργασία με διοικητικούς και προμηθευτές πρόσβαση στο ίντερνετ. Ιδού η νομική βάση της δράσης μας. Νόμοι για τις τηλεπικοινωνίες, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο ποινικό κώδικας και ο επίσης ποινικό κώδικας. Αυτά μας δίνουν τα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε το κυβερνοέγκλημα στην Πολωνία. Όλες οι οδηγίες της Ένωσης εφαρμόζονται επίσης. μια στιγμή δεν γυρίζει, ναι. Ειδού τι αναμένουμε τώρα για το μέλλον. Όλο και περισσότεροι τομείς της ζωής μας βασίζονται στον κυβερνοχώρο και θεωρούμε ότι ως αστυνομικοί πρέπει το νομικό σύστημα, το δικαστικό σύστημα να δίνει τη δυνατότητα για την πρόληψη εγκλημάτων και να επιτρέπει στις αρχές, στις ιδιοκτικές αρχές να δράσουν αποτελεσματικά με τη χρήση της τεχνολογίας που χρειάζεται καθώς και επαρκής κυρώσεις. Τώρα θα σας δείξω μερικές από τις κυριότερες περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει τον τελευταίο χρόνο. συμμετείχαμε στην καταπολέμηση ηλεκτρονικών ιών στο Πανεπιστήμιο το υλικό που χρησιμοποιήσαμε βασιζόταν και σε ευρωπαϊκή τεχνολογία 150 τερατομπάιτς χρησιμοποιήσαμε χώρου αποθήκευσης Επίσης, σε συνεργασία με το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών που εδρεύει στο ίδιο κτίριο, καταπολεμήσαμε, αποκαλύψαμε ότι υπήρχαν προσφορές δουλεμπορίου και εμπορίου εργάνων, οργάνων, ανθρωπίνων οργάνων. Πληροφορίες για 121 χρήστες που προσπαθούσαν να πουλήσουν όργανα ταυτιστήκαν από μας και οι πληροφορίες εστάλησαν στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών. Επίσης έχουμε μια ομάδα για τη συνεργασία με άλλα τμήματα της αστυνομίας και χάρη στις δραστηριότητες μας μπορέσαμε να βρούμε πληροφορίες στο ίντερνετ για τη διάδοση οδηγιών για την παραγωγή εκρηκτικών. Και αυτές οι πληροφορίες εστάλησαν στο κεντρικό γραφείο πληροφοριών και μπορέσαμε να στείλουμε στο δικαστήριο 22 χρήστες του Ιντερνετ. Από το 2006 συμμετείχαμε σε 30 διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης παιδικής πορνογραφίας και ως αποτέλεσμα 1380 χρήστες του ίντερνετ ταυτίστηκαν που διέδιδαν παιδική πορνογραφία και 365 από αυτούς εμινήθησαν. Για μας είναι πολύ σημαντικό ως αστυνομική αρχή να, να γνωρίζετε ότι και η Τράπεζα Δεδομένων που μας χορήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε πολύ χρήσιμη. Με τη βοήθειά της μπορέσαμε να ταυτίσουμε τους χρήστες αυτούς. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζαλεύσκη που μας ε, αναφέρατε την πολωνική εμπειρία και τώρα προτάσει της Προέδρου μας κυρίας Χολμάγερ θα ήθελα τα επόμενα 20 λεπτά να γίνει ο πρώτος γύρος ερωταπαντήσεων και σχολείων. Αν συμφωνείτε, τότε θα έλεγα να λέτε πρώτα το όνομά σας και να ονοματίζετε εκείνον προς τον οποίο θέτετε το ερώτημα. Ορίστε εσείς εκεί κάτω. Ανδρέας Μπράμς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοςδήποτε από τους ειδικούς σας απαντήσει. Μιλήσαμε για την σημασία που έχει η καταπολέμηση του εγκλήματο, αλλά εκτός από τον τελευταίο μιλητή δεν προσπαθήσαμε να το ορίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να οριστεί ανακατηγορία το κυβερνό έγκλημα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με τις κατηγορίες βέβαια. Υπάρχουν οικονομικά εγκλήματα, απάτες ή πωλήσει κλεμμένης περιουσίας βανδαλισμοί και ίσως και με μερικά πολιτικά εγκλήματα, άλλη κατηγορία η παιδοπορνογραφία και η δουλεμπορία και τρίτη κατηγορία η τρομοκουρατία. Ίσως ακόμα μια κατηγορία η, το λεγόμενο spyware και το εμπορικό σπάμ θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ. Έβδομη κατηγορία. Οι ιστοσελίδες καθεστώτων που δεν εγκρίνουμε. Ιράν, Βόρεια Κορέα κλπ. Δεν ξέρω αν έχουν ιστοσελίδες, αλλά αν έχουν θεωρούνται θεμητές ιστοσελίδες επιτρέπεται να, τους, να τις επισκέπτονται οι δυτικοί. Εγώ βέβαια δεν θα ήθελα αλλά εμποδίζομαι ή όχι. Α, πολύ ευρύ το ερώτημα, δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Μήπως ο κύριος Πουρατίνσκι. Η απάντησή μου δεν θα είναι ικανοποιητική, γιατί νομίζω ότι αυτό που παρουσιάσατε ε, είναι ουσιαστικά ε, θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, υπεράσπιση αυτών όσων λέγονται για την ασφαλεία στον κυβερνοχώρο. Εδώ εξετάζουμε κάποια δικήματα για τα οποία ε, τα οποία καλύπτονται από τον όρο επέθεση στον κυβερνοχώρο και έχουμε και μία ευρύτερη κατηγορία δικημάτων ε, που διευκολύνονται μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιείται το διαδικτύο ως εργαλείο δηλαδή. Και γι' αυτό ξέρετε η απάτη είναι πολύ παλιό ε, έγκλημα, αλλά το διαδίκτυο δίνει νέες διευρυμένες δυνατότητες διάπραξης απάτης. Το ίδιο ισχύει και για την κλοπή ταυτότητα. Ε, υπάρχει πριν την εφεύρεση του ίντερνετ, αλλά και πάλι το ίντερνετ δίνει νέε οδού. Τώρα δεν θα έλεγα τίποτα παραπάνω σε αυτό το στάδιο, γιατί νομίζω ότι ε, δίνουμε εδώ απλώς κάποιες κατευθύνες γραμμές. Ε, η Σύμβαση της Βουδαπέστης και του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, το στοχεύει κυρίως στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχουμε και μία σειρά άλλων αδικημάτων που σχετίζονται και με την παιδική πορνογραφία, το χάρη, που υπήρχαν πριν από το διαδίκτυο, αλλά διευκολύνονται από το διαδίκτυο. Τώρα, από τη σκοπιά της ε, ποινική νομοθεσία μα ενδιαφέρει να είμαστε αρκετά ακριβείς, έτσι ώστε να είναι σαφές ε, ποιες πράξεις θεωρούνται ποινικό δίκημα και ποιε όχι. Εσείς βασικά αναφέρετε κάποια θέματα που ίσως ε, είναι ουσιαστικά στο μετέχμιο του τι θεωρείται εγκληματικό και τι όχι. Μια άλλη κατηγορία που χρησιμοποιείται συχνά και σχετίζεται με τις ε, δραστηριότητες ε, που σχετίζονται με το Ιντερνετ της Κομισιόν είναι η διάκριση μεταξύ του παράνομου περιεχομένου και του επιβλαβούς περιεχομένου. Δηλαδή το παράνομο περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο νομοθέτησαν πρόσφατα, ακόμη όχι, δεν υπάρχει πλήρης υιοθέτηση ε, μιλώ για την οδηγία για την ποιοτική βιβλιογραφία, ενώ το επιβλαβέ περιεχόμενο είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος ε, να έχει μέτρα soft law, παραδείγματο χάρη υλικό επιβλαβέ για τα παιδιά και αυτό είναι... Και αυτός είναι σημαντικό τομέα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό έγκλημα ή κάτι παράνομο. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Κάποιος άλλος από το πάνελ, ο κύριος Μίλλερ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, πρέπει να ε, πούμε ότι αυτό που είναι ε, παράνομο εκτός του διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, παράνομο και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν αυτά τα δικήματα τα οποία αν διαπραχθούν οδηγούν σε μία κατάσχεση του υπολογιστή δεν μπορείς δηλαδή να, ε, ε, να επέμβεις παράνομα σε ένα άλλο ε, υπολογιστή σαν hacker. Αυτή τη διάκριση κάνουμε. Εγώ θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι ακόμη ότι ορισμένοι κυβερνοεγκληματίες είναι πολύ καλά οργανωμένοι και καλά εξοπλισμένοι ε, για να αναλάβουν πολύ περίπλοκες δραστηριότητες ε, ενδέχεται δεν είναι ε, πληρωμενοι και από τους τρομοκράτες. Η κυρία Χόλμαγερ τώρα. Έχω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά δεν έχει μικρόφωνο η ομιλήτρια. Έχω μία ερώτηση σχετικά με το χρονικό πλαίσιο της οδηγίας διότι εδώ αναφερόμαστε ε, σε θέματα τα οποία αλλάζουν καθημερινά άρα θα πρέπει να υπάρχει συνεχής αλλαγή Ακόμη λοιπόν και αν είναι πολύ ουδέτερη η διατύπωση της οδηγίας, τα προβλήματα που καλύπτει ε, θα αλλάζουν μορφή συνέχεια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο έχουν σκεφτεί η Προεδρία του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί ένας μόνιμος οργανισμός ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ε, συνεχώς ανανεωνόμενες προκλήσεις, διότι διαφορετικά θα πρέπει κανείς να προσέχει πώς θα ενημερώνει συνέχεια αυτή την οδηγία για να αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις των καιρών. Σας ευχαριστώ για αυτό το πολύ βασικό θέμα το οποίο είναι όντως ουσιαστικό. Κάποιος από εσά θέλει να απαντήσει. Η ε, Πολωνική Προεδρία. Θα προσπαθήσω. Σχετικά με την οδηγία πρέπει να σας πω ότι ήδη ένας από τους κανόνες τους οποίους ακολουθήσαμε στη συζήτηση στο Συμβούλιο είναι να έχουμε τεχνολογικά ουδέτερες διατάξεις, δηλαδή να καθορίζουμε ε, τις ιδέες του τι είναι το κυβερνοέγκλημα με ε, γενικές, γενικούς ορισμούς και να μην χρησιμοποιούμε ε, την τη γλώσσα των ε, τεχνικών αλλά να μπορούμε ε, πιο γενικά να γνωρίζουμε αν μία πράξη ε, εμπίπτει σε μία κατηγορία όντας αρκετά γενική ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε νέες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εγκληματίες αυτές για να τις καλύψουμε μέσω αυτής της οδηγίας. Αυτό είναι το κλειδί στο να υπάρχει ε, μια οδηγία που δεν χρειάζεται να ενημερώνεται ετησίως και αν μπορέσουμε να έχουμε τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να προβαίνουμε σε ε, αναθεωρήσεις τόσο συχνά. Ο κύριος Παρατίνσκι. Για να δώσω μια συνέχιση σε όσα υπόθηκαν. Νομίζω ότι είχαμε μια επιτυχή σύμβαση, την ε, Σύμβαση της Βουδαπέστης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θετήθηκε πριν 10 χρόνια. Και νομίζω ότι βασικά κατόρθωσε να επιβιώσει για να έχει νόημα λόγω της χρήσης ε, μη τεχνικά ουδέτερης γλώσσας. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και ορισμένες τροποποιήσεις. Έχουμε διατυπώσει το άρθρο 7 που μπορεί να διαβαστεί από πρακτική σκοπιά ως ένα μέτρο για να απαντήσουμε στις απειλές που δημιουργούνται από τα botnets, από τα δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ. Αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στο botnet αυτό καθ' αυτό. Δεν ε, περιγράφουμε εδώ, δεν έχουμε καμία τεχνική περιγραφή των τι είναι το botnet. Ε, που θεωρείται τώρα μία μείζον απειλή, μία μείζον απειλή. Ε, απλώς χρησιμοποιούμε δεύτερη γλώσσα όπως είναι εργαλείο, συσκευή, tool, device ή στο σημείο Β λέμε ε, παραδείγματο χάρη κωδικό πρόσβαση ε, κτλ. ή παρόμοια στοιχεία. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα ισχύει σε λίγα χρόνια. Ναι δεν ε, θα αποκλείσουμε ποτέ τη δυνατότητα κάτι να μας ξεφύγει από αυτούς τους ευρύς Αλλά μέχρι τώρα νομίζω ότι ήμασταν επιτυχείς. Και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι, αλλά φυσικά θα πρέπει να επαγρυπνούμε και νομίζω αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Έχω μια ερώτηση, λέει ο Το Σέλερ, που σχετίζεται με το σε ποιο επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα. Αν το δούμε από έξω, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκρεμεί μια νομοθεσία στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Προβλέπεται να υιοθετηθεί ε, και λένε ότι θέλουν να αρχίσουν διεθνείς διαπραγματεύσεις για την τυποποίηση, για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν πάλι πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη δομή, αλλά, με τη διάρθρωση, αλλά υπάρχει μεγάλη ευλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και του Κογκρέσου. Το κύριο ερώτημα όμω είναι, έπρεπε να μάθουμε αυτό το δείγμα όταν οι Αμερικανοί ε, άρχισαν ε, να αντιπαρατήθηκαν μαζί μας ε, για την ασφάλεια των κοντέινερ, των εμπορευματοκιβωτίων, όταν άρχισαν να μας ζητούν νομοθεσία. Και ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να φερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά διεθνείς και δημιουργικές διαπραγματεύσεις, παραδείγματος χάρη με τους Αμερικανούς για ένα τέτοιο ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν άμεσε επαφέ με του Αμερικανού και διάφοροι οργανισμοί όπω η Κομισιόν έχουν επαφέ με του Αμερικανού, αλλά για την, η νομοθεσία για την ασφάλεια των κοντέινερ Μα έδειξε ότι χρειαζόταν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διάρθρωση του διαλόγου. Ποια είναι η προσωπική σα άποψη Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα θέλουν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία οι Αμερικανοί, γιατί στην νομοθεσία λέει ότι μέσα σε ένα έτος πρέπει οι Αμερικανοί να το πράξουν αυτό, να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της πώς οργανώνεται για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα. Να ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις ε, από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και στη συνέχεια από τους υπολείπους ομιλητές. Δεν μπορώ να σας δώσω μία πλήρη απάντηση επί της ουσίας, καθώς αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο είναι αρμόδιοι συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Information Society, όμως επί της διαδικασίας. Νομίζω ότι κάναμε κάποια βήματα προς τα μπρος που θα μας βοηθούσαν να είμαστε πιο έτοιμοι. Ανέφερα την ομάδα εργασίας ε, των ΗΠΑ ε, για την ασφαλή στον χωρού και το κυβέρνο έγκλημα Εκεί θέλουμε να δυσκολήσουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για διευθετήσεις ad hoc ή για συναντήσεις ad hoc που ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά υπάρχει μία συνέχεια. Και υπάρχει η πρόθεση στην επόμενη Σύνοδο Κορφής με τη να συστήσουμε ε, την δημιουργία κάτι τέτοιου, ενός τέτοιου οργάνου. Όπως σας είπα, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Σε εσωτερικό επίπεδο, και νομίζω ότι το έφερε αυτό και συνάδελφος από την Εσθονία, δηλαδή ως προς τον εσωτερικό συντονισμό, και πάλι κάναμε κάποια βήματα πριν λίγους μήνες, αρχή ξεκινήσαμε ε, συναντήσεις στα πλαίσια μιας διαπηρεσιακής ομάδας ε, όπου συμμετέχουν διάφορες υπηρεσίες κομισιών ε, και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης για να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον είμαστε καλά ενημερωμένοι σε σχέση με το τι κάνουν τα διάφορα μέρη. Και δημιουργείται και ένα πεδίο για συντονισμό. Δηλαδή, αυτή είναι κάποια εσωτερική δουλειά που ξέρουμε ότι έπρεπε να την κάνουμε και μας βοηθά να έχουμε μια πιο ενοποιημένη απάντηση και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση συντονίζει την ομάδα αυτή. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, κύριε κλάση. Νομίζω ότι σχετικά ε, με αυτήν την ε, νομοθεσία που διατύπωσε το Κογκρέσο είναι δύσκολο να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο κατερτισμένη από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σχετικά με την προστασία του ατόμου ε, και σε παρεμφερείς τομείς. Πολλές φορές ε, δεν ε, γίνεται κατανοητό ότι δεν είμαστε ένα ομόσπονδο σύστημα διότι εμείς δεν έχουμε λευκό ήχο και δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε στις πρωτεύουσε, τι θα κάνουν. Οπότε νομίζω ότι στο μέλλον θα βλέπουμε όλο και περισσότερο να ζητούν, να αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μία οντότητα σε διάφορους τομείς. Οπότε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί και να αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σαν μία ενιαία μονάδα είτε πρόκειται για το κυβερνοέγκλημα είτε για άλλους τομείς. Ωραία. Λοιπόν, Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεργαστήκαμε ε, ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να σχολιάσει σε αυτό το σημείο. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή την νομοθεσία, αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε στα προβλήματα αυτά και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με τις Ηνωμένε Πολιτείες και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα καταπολεμά τους ίδιους στόχους. Ε, λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση από πίσω. κάποιο σήκωσε το χέρι του. Μπορείτε παρακαλώ να πείτε το όνομά σας. Είμαι μία δημοσιογράφος από το Observer. Ε, θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται ε, σχετικά με αυτή την οδηγία Εάν εξετάζουμε και τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως στην Ολλανδία το DG Notar που εξέδωσε πλαστά πιστοποιητικά που έμοιαζαν σαν Google ή μηνύματα ηλεκτρονικά για κατασκοπία του Ιράν και τα λοιπά. Ε, ε, βέβαια εντωμεταξύ έκλεισε αυτό το σύστημα η κυβέρνηση της Ολλανδίας αλλά ε, ήταν δυσάρεστο και πώς θα αποφύγει κανείς να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι περιγράψατε αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, δεν ασχολούμεθα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ε, οπότε δεν ξέρω τι έκανε κάποια εταιρεία και αν αυτές οι πράξεις είναι, ε, θεωρούνται αξιόπινες σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Ε, όσον αφορά τη, τις εγκληματικές ενέργειες ε, βεβαίως θα επεμβαίναμε αλλά όσο προς τα τεχνικά στοιχεία δεν μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ. Τώρα είναι, έφτασε η ώρα να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος και δίνω το λόγο και πάλι στην κυρία Χολμάγερ. Προσπαθώ να βρω πού είναι τα μέλη του, της, ε, για το δεύτερο μέρος Μπορώ να ξεκινήσω την εισαγωγή ε, σχετικά με το δεύτερο μέρος εφόσον ήρθαν οι συμμετέχοντες και εδώ ε, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας πούν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα. Βλέπουμε τον κύριο Χάντζο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Σίμαντεκ, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι ε, μας ε, είπε διάφορα ανέκδοτα που βλέπει κανείς στο διαδίκτυο και επίσης έχουμε αυτούς όπου υπάρχουν οι τα μεγαλύτερα προβλήματα και ε, γι' αυτό βλέπω ότι εκτός από τους, τον εκπρόσωπο της Γερμανικής Ένωσης Τραπεζών έχουμε έναν εκπρόσωπο του Chaos Computer Club στη Γερμανία ο οποίος θα μας πει πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα άρα σας καλωσορίζω και δίνω πρώτα τον λόγο στον κύριο Χάντζο. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές που έδραξαν την ευκαιρία να οργανώσουν αυτή την ακρόαση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και που μου δίνουν τη τιμή να απευθυνθώ εδώ σήμερα σε εσά. Έχουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Πρέπει να συζητήσουμε ποιο είναι ο ρόλο του ιδιωτικού τομέα και τι μπορεί να γίνει για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματο και την πρόληψή του. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό από τη σκοπιά της ε, Semantic, καθώς είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, εταιρείε ε, που παρέχει υπηρεσίε για τις κυβερνήσεις, για τους καταναλωτές, για την ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητούμε τη κυβερνοαπειλή και όταν συζητούμε την εξέλιξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε πώς έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, τι πρέπει να αναμένουμε όταν ε, συζητούμε το πού πάει η τεχνολογία. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε ε, σε ένα σημείο ε, ε ιστορικά οι τεχνολογίες, ο τρόπος που οργανώνουμε τις τεχνολογίες των πληροφοριών επικεντρώνονταν στο σύστημα, βασίζονταν στο hardware, στο λογισμικό ε, και υπήρχε πολύ μεγάλος έλεγχος ενώ τώρα απομακρυνόμαστε από αυτό σε μια προσέγγιση που βασίζεται στις πληροφορίες που επικεντρώνεται στις πληροφορίες δηλαδή είναι τα δεδομένα που έχουν πλέον αξία όχι ε, το hardware και οι πληροφορίες είναι το αίμα της κάθε επιχείρησης χρησιμοποιούμε το cloud computing ε, και την ε, σε εικονικές τεχνολογίες, virtualization. Ε, επίσης, νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά γεγονότα σε σχέση με το κυβερνό έγκλημα και αυτά που σας παρουσιάζω σήμερα, ή τα νούμερα, προέρχονται από μια έκθεση που δημοσιεύσαμε πρόσφατα σε σχέση με την πλήρη κλίμακα του κυβερνού Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και σε βασική έρευνα που κάναμε σε πολλές χώρες γύρω από τον κόσμο. Καταρχήν, βλέπουμε ότι το άμεσο κόστος της μετρητής, ε, δηλαδή τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί ή έχουν κλαπεί φτάνουν τα 114 δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, η, μαύρη αγορά ε, των ε, όσων ε, έχουν κλαπεί ουσιαστικά ανταγωνίζεται την αγορά των ναρκωτικών. Αν ε, συγκρίνετε μπορεί να φτάσετε το χάρη 100 φορές των ετησίων δαπανών της UNICEF και επίσης το το 10% των ενηλίκων έχουν βιώσει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στο κινητό τους. Έτσι λοιπόν ιστορικά θεωρούσαμε το κλίμα στον κυβερνοχώρο ως μία πτυχή απειλής ε, στα κέντρα δεδομένων και στους προσωπικούς υπολογιστές. Τώρα γίνεται όλο ένα και περισσότερο ένα στοιχείο που ε, πλήττει και τα κινητά μας και όσο πιο έξυπνα τα κινητά μας ε, τόσο περισσότερο θα δέχονται επιθάσεις. Πέρσι, σε 24 χώρε, 431 εκατομμύρια ενηλικέ βίωσαν έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο ήταν θύματα σε καθημερινή βάση. Και αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για 14 ενήλικε το δευτερόλεπτο. Τώρα, αν ε, μίλησα για την εξέλιξη των ε, τεχνολογιών της πληροφορικής, κινητικότητα, cloud computing, έχουμε ε, έκρηξη του αριθμού των πληροφοριών που παράγουμε. Είπα ότι πέρσι παρηγάγαμε 380 ε, δισεκατομμύρια DVD. Αυτά είναι όλα τα δεδομένα που είναι και έξω στο ίντερνετ και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε διπλασιάσει αυτό το νούμερο. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η αίθουσα είναι πλήρως γεμάτη με DVD και πάλι δεν θα φτάναμε στον ε, αριθμό που έχουμε και έξω. Έτσι λοιπόν ε, πάρα πολλές πληροφορίες ε, ε, παράγονται. Έχουμε το cloud computing και την κινητικότητα και έχουμε και ένα αυξανόμενο και επίμονο αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να τονίσουμε τις λεγόμενες targeted attacks, στοχευμένες δηλαδή, επιθέσεις που έχουν ως στόχο στο να θέσουν σε κίνδυνο μία υποδομή καθώς είναι μοναδικές στο σχεδιασμό τους και είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέψουν στον επιτιθέμενο ε, μάλλον σε αυτόν που επιτίθεται, ε, να σκλέψει τις πληροφορίες ε, και να φύγει χωρίς να τον βρουν. Έχουμε επιθέσεις όπως το Stuxnet και άλλες και πρόκειται για ονόματα που ακούσαμε το 2010 πολλές φορές. Άλλη απειλή που είδαμε είναι της κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα το ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα ως αποτέλεσμα αυτό Νομίζω ότι ε, αν ε, συγκρίναμε το Facebook με μια χώρα θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν σε τέτοια περιβάλλοντα ανθεί το κυβερνό έγκλημα και προσπαθούν ε, ε όσοι επιτίθενται να βελτιώσουν τις τεχνικές τους, προσπαθούν να βρουν ευάλωτα σημεία που δεν έχουν εντοπιστεί και υπάρχει επίσης και εκδημοκρατισμός των επιθέσεων. Δηλαδή υπάρχουν εκεί έξω εργαλεία που καθένας από εμά μπορεί να αγοράσει online ε, και να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει μια επίθεση. Έτσι, ε, λοιπόν, αν δούμε τις 10 κύριες χώρες όπου έχουμε συνήθως κακόβουλη, από τις οποίες συνήθως προέρχεται η κακόβουλη δραστηριότητα, βλέπουμε και την Κίνα και για αυτή θα σας μιλήσω. Πολύ συχνά μιλάμε για την Κίνα ότι είναι μεγάλη πηγή κυβέρνο επιθέσεων προς τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας εκπλήσει ότι χώρες όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σημαντική αναλογία και δεν μας εκπλήσει γιατί έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό αλλά και πολύ μεγάλη δίσδυση ευρυζωνική. Αλλά αν προσθέσετε τρει χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία, σε αυτή την περίπτωση σχεδόν φτάνετε στα ποσοστά τη Κίνα. Δηλαδή τι προσπαθώ να πω εδώ, ότι υπάρχει πολύ έγκλημα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και σημαντική παρουσία της δραστηριότητας στο εσωτερικό της Ένωσης και πρέπει να θυμόμαστε κάτι πολύ σημαντικό στα στατιστικά στοιχεία. Η κακόβουλη δραστηριότητα αναχώρα δεν υπονοεί ότι προέρχονται οι επιθέσεις από εκεί, δηλαδή ότι βασίζονται ε, όσοι επιτίθενται οι δράστε σε αυτές τις χώρες, αλλά χρησιμοποιούν εκείνου του υπολογιστέ σε εκείνε τι χώρες. Αυτοί οι υπολογιστέ είναι το τελευταίο σημείο από το οποίο περνούν οι δράστε πριν να ξεκινήσει η επίθεση. Δηλαδή αυτό δεν μα λέει που μένουν οι hacker, που βρίσκονται, απλώς ε, μας λένε ότι προέρχονται οι επιθέσεις από αυτά τα περιβάλλοντα. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική και βλέπετε τι πολίτες στο διαδίκτυο και πόσο και πόσο κοστίζουν. Προφανώς ε, οι δράστες ε, θέλουν τις χρηματοπιστικές πληροφορίες ε, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τις πιστοτικές και οι λογαριασμοί email επίσης τους ενδιαφέρουν. Επίσης έχουμε παραβιάσει ασφαλεία. είμαστε στη μία την εβδομάδα, συνεχίζουν να έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο κατά μέσο όρο. Έχουμε 260.000 ε, ταυτότητες που αποκαλύπτονται ανά παράβαση και βλέπουμε ότι το μέσο κόστος ε, είναι πολύ πιο ψηλό ε, από ότι μπορεί να έχουμε το χάρη από την τυχαία απώλεια ή ε, τη μη ασφαλή πολιτική. Έτσι λοιπόν οι δράστες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί όταν έχουμε εξωτερική επίθεση. Ένα μέσο κόστος για να επιληθεί μια τέτοια επίθεση κατά των δεδομένων δεδομένων είναι 7,2 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή έχουμε και πάλι κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο στόχος γίνεται οι πληροφορίες, όχι απαραίτητα υποδομές. Και μιλήσα, μίλησαν οι συνάδελφοι για την Εστονία, και για άλλα κράτη βλέπουμε στόχοι να είναι περισσότερο κυβερνήσεις και κυβερνητικές ε, υποδομές. Αυτό είναι πολύ αισθητικό για πολλούς λόγους. Γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να ε, προέρχεται στο ότι οι κυβερνήσεις έχουν πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, στοιχεία, πολύτιμα και επίσης ε, το ότι Παραδείγματο χάρη, μια επιτυχής ε, επίθεση μπορεί να ξεκινήσει από ένα κυβερνητικό ε, όργανο. Έτσι λοιπόν είναι αυτό ένα φαινόμενο που αρχίζουμε να βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και στο μέλλον. Τώρα, κριτική υποδομή και αυτή έχει δεκτεί επίθεση. Πολύ. Ε, ε ε, την επίθεση κατά των ε, Ιρανών πυρανικών, Ιρανικών πυρονικών υποδομών ως κάτι που τους ε, ξύπνησε με το Stuxnet, όμως κάτι που έκανε το Stuxnet πιο αποκαλυπτικό από άλλα ήταν ότι το Stuxnet ήταν μια επίθεση που είχε ουσιαστικά ένα φυσικό αποτέλεσμα, δηλαδή να σεμποτάρει την υποδομή. Ποτέ δεν είχαμε βιώσει κάτι τέτοιο, τέτοια ικανότητα ε, και νομίζω ότι εδώ βλέπουμε μια μεγάλη αλλαγή προ αυτή την κατεύθυνση. Όμω αυτή δεν ήταν η μόνη περίπτωση και οι στατιστικέ μα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η τόση. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι ο ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Άλλοι το είπαν επίση. Η άποψή μα θα ήταν ότι το έγκλημα στην κυβερνοχώρα δεν μπορεί να επιληθεί μόνο από μια κυβέρνηση σε μια χώρα. Η ε, πραγματικότητα επίση είναι ότι η υποδομή των ε, τεχνολογιών είναι κυρίως στα χέρια του ιδιωτικού τομέα χρειάζεται μία συλλογική προσέγγιση και μία συλλογική άμυνα όπως γίνεται στο ΝΑΤΟ. Ο ιδιωτικός τομέας έχει συμφερόν να αναπτύξει ε, υποδομές ασφαλής και αναπτύξει την τεχνολογία για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Αυτό πράττουμε ταυτόχρονα Πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τεχνολογικές πληροφορίες και ασφάλεια δεν είναι οι μόνες λύσεις. Ναι. Ε, μιλάμε για μια ομάδα εδώ και νομίζω ότι οι χαράκτες πολιτικές πρέπει να αναπτύξουν ε, ένα εύρωστο νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχει φυσικά και ε, μια προσωπική απευθυνότητα. Ε, και το ερώτημα είναι τι γίνεται με την αξιολόγηση κινδύνου. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνουμε τι κίνδυνο διατρέχουμε και ποιο επίπεδο ασφάλεια πρέπει να έχουμε έναντι αυτού του κινδύνου, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα αποτελεσματικά. Και κλείνοντα τι πιστεύουμε για τη σημερινή πρόταση. Να πούμε ότι είναι ρεαλιστική ως προς το πεδίο εφαρμογής και τις δυνατότητες για κατάληξη συμφωνία. Αν δω το παρελθόν, ε, είχαμε ε, μία διαπραγμάτευση και είχαμε και την απόφαση ε, πλαίσιο για το έγκλημα στην χώρο. Αυτό θέλει να τροποποιήσει η σημερινή πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε ίσως να συζητήσουμε το θέμα των επιβαρυντικών περιστάσεων που μπορούμε να έχουμε κάτι πιο ισχυρό σε ποιους τομείς, αλλά η σημερινή πρόταση οδεύει προς την κατεύθυνση δεν ε, μπορούν να καλυφθούν όλες οι μορφές εγκλήματο στον κοινωνικό χώρο. Τώρα για τις στάσεις στο μέλλον θα σας ε, καλώς σκεφτείτε την κλοπή ταυτότητας καταρχήν και την ε, απάτη μέσω υπολογιστή ε, συζητούνται αυτά και στη Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης, κλοπή πληροφοριών. Πολλοί αναφέρθηκαν ε, στην, στην κλοπή προσωπικών δεδομένων, αλλά τι γίνεται με την πνευματική διοκτησία. Επίσης, ε, αναφέρθηκε και το θέμα της κλοπής των πόρων, ε, ε, δηλαδή κάποιοι χρησιμοποιούν το cloud computing χωρίς δικαίωμα και επίσης έχουμε και τις πτυχές του δικονομικού δικαίου που καλύπτεται από τη Σύμβαση του, Ευρωπαϊκού, συγγνώμη, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ να απαντήσω ερωτήσει. Ευχαριστώ κύριε Χάντσο και τώρα δίνω το λόγο εις ε, τον κύριο Βάλτερμαν Γκούτσιν και του δίνω αμέσως τον λόγο. Προσπαθεί βέβαια προς το παρόν να ε, δει πώς ε, θα χρησιμοποιήσει ε, το λάπτοπ του. Θα μιλήσω γερμανικά γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα. Εργάζομαι επί 10 χρόνια στον τομέα της ασφαλείας για τον κωδικό PIN στις γερμανικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν μία σημαντική ε, αύξηση των επιθέσεων της ε, κυβερνοεγκληματικότητες στις ε, διάφορες δομές και του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού και βλέπουμε ότι υπάρχουν τα ΣΠΑΜ, τα DDoS και αυτά ιδίως πλήττουν τις τράπεζες και τώρα έχουμε ε, και τα botnets τα οποία είναι σημαντικό εργαλείο για αυτές τις επιθέσεις ε, σε μία ερώτηση μίας ε, δημοσιογράφου αν θα ε, σταματήσει η DG Notar βεβαίως και θα συνεχίσει να λειτουργεί ε, αλλά βλέπουμε την Sony, βλέπουμε την RSA η οποία έχει ε, τον υπολογιστό στη Linux και ξέρουμε τι έχει τραβήξει η DG Notar όπου και πάλι ο υπολογιστής ήταν Linux για την Notar στην Ολλανδία. Και πάντοτε υπάρχουν δημοσιεύσεις, επικεφαλίδες, πρώτες σελίδες στην εφημερίδα ε, και ε, υπάρχει και το Miner Botnet το οποίο ως επτοπλίστων ε, είναι κάτι το οποίο δεν καταρτίζεται στη Γερμανία αλλά χρησιμοποιείται στη Γερμανία. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από επιθέσεις της σημερινής εποχής και λάθη τα οποία συμβαίνουν παρόλα τα πιστοποιητικά και παρόλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει αυτή η οδηγία θα συνεχίσουν. Ε, έχουμε ιδίω στον ε, τομέα της ε, πίστεως και των τραπεζών διάφορα προβλήματα και όπως είπε εδώ προλαλή σας, βλέπουμε ότι έχουμε 500, ε, ε, ε, από, 5.000 μέχρι 500.000 περιπτώσεις τρόγιαν, τροικών δουλειών ύπων στη Γερμανία και βλέπουμε ότι μπορεί να είμαστε σε έναν πιο καλό κόσμο αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Πολύ σύντομα λοιπόν πρέπει να είμαστε συνέχεια σε γρήγορση και να προσπαθούμε να βελτιωθούμε και στη Γερμανία από το 1990 έχουμε πλέον αυτή την identification με δύο παράγοντες και έχουμε διάφορα πρότυπα τα οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε όπως ε, είναι Digital Signature, Index TAN, Mobile TAN, Chip TAN και ακόμη και Photo TAN το οποίο ε, ετοιμάζεται τώρα. Τελικά όμως ε, όλη η τεχνική είναι πάνω στο τσιπάκι που είναι πάνω στην κάρτα. Μέσω αυτού μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε και την εγρήγορση των χρηστών. Έχω εδώ ένα αφιλάδιο το οποίο ίσως μπορείτε να διαβάσετε, αλλά ουσιαστικά όπως σας είπα τα δύο βασικά σημεία είναι ε, το τσιπάκι και ο άνθρωπος. Μερικά παραδείγματα. Βλέπετε εδώ το, ε, διάφορες το φωτοτάν, το best sign και το chip tan ε, το φωτοτάν είναι τη μίας τράπεζας της Commerzbank και υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις τις οποίες προωθούμε. Και εμείς χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ένα πρώτο βήμα αλλά ένα επιτυχές δεύτερο τρίτο βήμα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια διότι υπάρχει μεγάλη απειλή για την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη και αυτό προσπαθούμε και εμείς να ε, λύσουμε ιδίως όταν πρόκειται για εγκληματικούς στόχους και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την οδηγία αλλά και η βιομηχανία και το κράτος πρέπει να μπορεί να προστατευτεί, να αναπτύξει αντίμετρα και ε, να μπορέσει ε, να προχωρήσει γι' αυτό και έχω διατυπώσει την ε, πρότασή μου. Δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο στην τεχνική αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός διότι μπορεί οι ε, τράπεζες ε, να μπορούν ε, να αντεπεξέλθουν αλλά βλέπουμε ότι οι εγκληματίες δεν επιτίθενται μόνο στις τράπεζες αλλά και σε άλλες δομές είτε πολιτικές είτε εμπορικές όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως πρόσβαση σε ανηλίκους και δεν είναι δηλαδή ο μόνος στόχος οι τράπεζες και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σωστό πλαίσιο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ε, ε, να καταρτήσουμε τις αναγκαίες δομές. Και ε, ολοκληρώνω την παρουσίασή μου πρέπει να υπάρχει συνεργασία των ε, EISPs για να μπορέσουμε να προλάβουμε και ε, να καταστήλουμε τις ε, αξιόπινες πράξεις και να εμποδίσουμε και να διώξουμε τα ISPs που προσπαθούν να απορρίψουν ή να εμποδίσουν τα μέτρα αμήνης. Ε, χρειάζεται καλύτερη και γρηγορότερη διασυνοριακή συνεργασία, ανάπτυξη καλών υποδομών και στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που πρέπει να ξεκινήσουν. Δεν ε, υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία ε, να μπορέσει κανείς να θεωρήσει ότι θα λύσει το πρόβλημά του μόνος του. Και υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις χώρες όπως οι Ηνωμένε στην Ευρώπη ε, που προχωρούν η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία ε, και θα μπορέσουμε ίσως ε, να καταρτήσουμε μια ενιαία στρατηγική καταπολεμήσεως του κυβερνοεγκλήματος με τρόπο στοχευμένο και με μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να διευρύνουν τη χρήση των μηχανισμών που διαθέτουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ για την γρήγορη αυτή επισκόπηση και τώρα θα κάνουμε μία αλλαγή στο λογισμικό του λάπτοπ.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 So, jetzt Λοιπόν, και με μεγάλη χαρά χαίρομαι ότι είναι εδώ ο κύριος Βάλτερ, ο οποίος θα μας δώσει μια διαφορετική οπτική γωνία στα θέματά μας και γι' αυτό και χαίρομαι, ναι. Τουλάχιστον προσπάθησα να σας παρουσιάσω μια διαφορετική οπτική γωνία, διότι θα μιλήσουμε για το κυβερνοέγκλημα από την σκοπιά του επαγγελματία hacker. Τώρα βρίσκομαι στο τέλος, άρα Σύντομα, σύντομα λοιπόν, να σας, πω ποιος, να σας πω ποιος είμαι. Είμαι επαγγελματίας Χάκερ από το 99. Έχω εργαστεί σε διάφορους consultant διεθνείς. Έχω μία δεκαετία εμπειρίας με εταιρείε και κυβερνητικά ηλεκτρονικά συστήματα από μέσα και από έξω. Τα ξέρω όλα αυτά. Ήμουν μέσα, γνωρίζω τα συνθήματα, έχω μπει μέσα και ένομα και παράνομα. Μερικά γενικά. ποια είναι η ρίζα του προβλήματος εδώ. Το πρόβλημα είναι το κυβερνοέγκλημα, έτσι. Λοιπόν λοιπόν. Γιατί αυξάνεται ενώ όλα τα άλλα είδη εγκλημάτων μειώνονται. Το σκεφτήκατε ποτέ. Είναι γιατί είναι κάτι απλό, εύκολο, με περισσότερο κέρδος και λιγότερο κίνδυνο από ότι τα υπόλοιπα είδη εγκλημάτων. Είναι ευκολότερο να μπει κανείς μέσα σε μια τράπεζα ηλεκτρονικά από ότι, μια, από ότι πραγματικά και από ένα χολτά μπορεί να πάρετε 5-10 χιλιάδες ευρώ ενώ ηλεκτρονικά εκατομμύρια. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το κυβερνοέγκλημα και αυξάνεται αντί να μειώνεται όπως τα περισσότερα άλλα είδη εγκλημάτων στον κόσμο. Γιατί όμως είναι τόσο εύκολο και ελκυστικό για τους εγκληματίες. Διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να το αντιμετωπίσει αυτοί που πουλούν software δεν ενδιαφέρονται να είναι και ασφαλές. Οι εταιρείε τι υπογράφουν όταν δημιουργούν ένα σύστημα. Digital passport, έτσι το λένε, αλλά αυτό δεν διασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος. Και υπάρχουν λάθη που είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Έχω εδώ το σύνθημα μιας γνωστής εταιρείας ήταν prod admin από το production administrator. Πολύ εύκολο να το φανταστεί κανείς. Ολόκληρο το σύστημα λοιπόν ήταν λανθασμένο από την αρχή και δεν ακολουθούσε καν τις στάνταρ συμβουλές. Αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δίνονται εγγυήσει για την ασφάλεια ενός προγράμματος software, ενός προϊόντος software. Για τα αυτοκίνητα υπάρχουν εγγυήσει και είναι και πολύ ακριβές για τον κατασκευαστή. Ενώ πουλάει κανείς software που δεν δουλεύει από πλευράς ασφαλείας τι γίνεται, τίποτε απολύτως. Το software γράφει ότι, είναι ως, ότι πωλείται ως έχει χωρίς εγγύηση. Είναι η πρώτη φράση όλων των αδειών software στον κόσμο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους η παραγωγή software χωρίς εγγύηση. Γιατί. Αυτό πρέπει να αλλάξει και γι' αυτό πρέπει ο κίνδυνος να ε- μετακυλιστεί στον παραγωγό. Άμα του κοστίζει χρήματα τότε θα το προσέξει. Και έτσι θα πάψει να αυξάνεται κατά 80% περίπου το κυβερνοέγκλημα. Οι διαχειριστές των ηλεκτρονικών συστημάτων, δημιουργούν ηλεκτρονικά διαβατήρια όπως λένε, αλλά δεν το κάνουν όπως πρέπει. Διασυνδέουν όλα τους τα δίκτυα με ένα κεντρικό και άμα κανείς μπει στο κεντρικό τα βλέπει όλα. Αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος. Είναι ανοησία. Και είναι ακόμη πιο ανόητο να υπογράφει κανείς τα ηλεκτρονικά του διαβατήρια. Δεν γνωρίζω μία μόνο περίπτωση που γίνεται αυτό πολύ εύκολα και το έχω δει παντού από κατασκευαστές αυτοκινήτων μέχρι τράπεζες. Και των περισσότερων το βασικό σύνθημα λεγόταν root, admin ή secret one, two, three, γελία συνθήματα δηλαδή. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Άρθρα 3 με 6. Εδώ θα ήθελα να διαγραφούν, να διαγραφούν απλώς. Διότι αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι κάποιο σύστημα δεν είναι ασφαλές, δεν πρέπει να τιμωρείται αυτός που το απέδειξε, αλλά αυτός που μας είπε ότι το σύστημα είναι ασφαλές, ενώ δεν ήταν. Πρέπει να τιμωρείται αυτός που πουλάει συστήματα ασφαλείας που δεν είναι ασφαλή. όχι τον διαχειριστή, που, τον διαχειριστή που έβαλε σύνθημα αυτό που σας έλεγα πριν Secret αν του three, κάτι τόσο γελίο. Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα περισσότερα συστήματα είναι πολύ ευάλωτα. Άρθρο 6. οι ηλεκτρονικές εκπομπές, οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές δεν πρέπει να τιμωρούνται γιατί αν πάρετε όλα σας τα μυστικά έγγραφα στο σπίτι και τα πετάξετε από τον μπαλκόνι το λογαριασμό σας, το διαβατήριό σας, το πιστοποιητικό γεννήσεως, τα πετάξετε όλα και κάποιος στο δρόμο τα πάρει και τα διαβάσει και ξέρει πότε γεννηθήκατε και πού και πού είναι ο λογαριασμός σας κτλ. Ποιος πρέπει να τιμωρηθεί, αυτός που βρήκε τα χαρτιά στο δρόμο και τα διάβασε ή αυτός που τα πέταξε από τον μπαλκόνι. Νομίζω αυτός που τα πέταξε από τον μπαλκόνι πρέπει να τιμωρείται, όχι εκείνος που τα βρήκε και τα διάβασε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τι θα γίνει οι κατασκευαστές των συστημάτων δεν ενδιαφέρονται. Πρόκειται για συστήματα όντως που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα και κάποιος φυσικά θα τα πάρει, θα τα λάβει. Όλα τα προβλήματα αρχίζουν με τη φράση «κανείς δεν θα τολμούσε να και όμως θα τολμούσε». Άρθρο να διαγραφεί. Είναι τελείως ανόητο και με συγχωρείτε που το λέω έτσι, είναι βλακώδες. Θέστε δύο απλά ερωτήματα. Αν χάσετε τα κλειδιά του σπιτιού σας, τι κάνετε. Δημιουργείτε νομοσχέδιο που κάνει, θεοκαταστά, καθιστά παράνομη την απώλεια κλειδιών ή αλλάζετε την κλειδαριά. Εγώ θα άλλαζα την κλειδαριά. Αν αλλάξετε την κλειδαριά, τότε δεν έχει νόημα ποιος έχει τα παλιά κλειδιά διότι δεν θα μπορεί να ανοίξει την πόρτα. Άμα αντιδράει κανείς σωστά δεν χρειάζεται να νομοθετεί αχρήστος. Τώρα οι αυξημένες κυρώσεις. Υπάρχουν αυξημένες κυρώσεις για τα κυβερνοεγκλήματα και άλλα εγκλήματα όλο και περισσότερες εδώ και μερικά χρόνια από τη 11η Σεπτεμβρίου βασικά. Αλλά έχουμε δει λόγω των αυξημένων κυρώσεων να μειώνεται το κυβερνοέγκλημα. Είναι λιγότερο. Όχι. Περισσότερο. Και γιατί είναι περισσότερο αφού αυξήσαμε τις κυρώσεις. Μήπως γιατί η αύξηση κυρώσεων δεν βοηθάει καθόλου. Έτσι νομίζω. Άρθρο 8. Η δημοσίευση ευαίσθητων στοιχείων είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι αν θέλουμε να προστατέψουμε τα συστήματά μας πρέπει να ξέρουμε τι προστατεύουμε. Αν δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος τότε δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο αν όχι αδύνατο να το προστατέψουμε αποτελεσματικά. Το να γίνεται παράνομη η δημοσίευση πληροφοριών για τα αδύνατα σημεία συστημάτων υποδομών και software μας μειώνει την ασφάλεια γιατί οποιοδήποτε έχει αυτές τις πληροφορίες μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ενώ εμείς που δεν τις έχουμε δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει ο κίνδυνος και γι' αυτό δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Λύστε το και αυτό λοιπόν παρακαλώ. Αν και η απλή δοκιμή των αδυναμιών είναι έγκλημα, τότε κανείς δεν θα δοκιμάσει. Αλλά είναι ουσιώδες για μας αν ένας 14χρονος Βραζιλιανός προσπαθήσει να μπει στο σερβερ του email της Κομισιόν και το καταφέρει, καλύτερα να το μάθουμε. Αν δεν το ξέρουμε, τότε ο 14χρονος Βραζιλιανός μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά του και δεν θα το ξέρουμε καν. Άρθρο 9. Το ίδιο με αυτό που είχα πει πριν, έχουν αυξηθεί οι κυρώσεις πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν βλέπουμε καμία μείωση του εγκλήματος. Γιατί να τις αυξήσουμε παραπάνω, δεν βοηθάει αυτό. Άρθρο 10. Το άρθρο 10 είναι το πιο γελίο από όλο αυτό το έγγραφο. Τα αναποδογυρίζει όλα θα έλεγα να διαγραφεί τελείως. Στην παράγραφο 1, η παράγραφος 1 θα έπρεπε να ονομάζεται η ανώνυμη παράγραφος, γιατί δεν έχει ως στόχο παρά μόνο να κατηγορήσει, να καταδικάσει ανώνυμους ανθρώπους. Δεύτερον, οι επιπτώσεις μιας επίθεσης. Λέει ότι πρέπει να τιμωρείται κανείς περισσότερο αν είναι σοβαρότερη η ζημιά. Τι ορίζει όμως την επίπτωση μιας επίθεσης. Αφού είπαμε ότι υπάρχουν για μεγαλύτερη ασφάλεια χωριστά κομμάτια ενός συστήματος για να είναι λιγότερο αποτελεσματική η επίθεση, για να είναι η ζημιά το δυνατόν μικρότερη. Αν κάποιος δεν το κάνει γιατί θέλει το σύστημά του να είναι πιο εύκολο, πιο απλό και φτηνότερο, τότε θα έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες και ζημιά αν υπάρξει επίθεση. Ο επιτιθέμενος λοιπόν τιμωρείται επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά του ο διαχειριστής. Δεν μου φαίνεται ούτε αυτό σωστό. Εάν ο διαχειριστής κάνει λάθος τη δουλειά του εκείνον να τιμωρήσετε. Αλλά τον να τιμωρείται κάποιος άλλος αντί από τον διαχειριστή δεν έχει νόημα. Τώρα η κλοπή ταυτοτήτων. Αναρωτηθείτε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση στις κλοπές ταυτοτήτων το ίδιο με αυτό που είπαμε πριν, γιατί είναι εύκολο, γρήγορο και αποδοτικό και με πολύ λιγότερους κινδύνους. Γιατί είναι τόσο εύκολο όμως. Γιατί έχουμε συνεχώς και περισσότερες τεράστιες τράπεζες δεδομένων με ευαίσθητα στοιχεία που απαιτούνται από ανόητους νόμους. Και υπάρχουν αυτά τα τεράστια ποσοστά στοιχείων στο ίντερνετ, τεράστιες τράπεζες δεδομένων που δεν αναζητούν, που δεν εφαρμόζονται με την δέουσα ασφάλεια. Αν υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα για 500.000 ε, κατοίκους της Ευρώπης θα βρεθεί κάποιος hacker να μπει μέσα. Γιατί, γιατί τον ενδιαφέρει να κλέψει 500.000 ανθρώπους. Αυτό είναι, έχει το μεγαλύτερο κέρδος και είναι και λίγη δουλειά. Είναι πολύ ευκολότερο να μπει κανείς κρυφά σε αυτή την τράπεζα δεδομένων παρά σε 10 μικρότερες. Αν δεν σταματήσουμε τη συσσόρευση αυτή τεράστιων ποσοτήτων στοιχείων σε μία τράπεζα δεδομένων δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλοπές των ταυτοτήτων. Θα συνεχίσουν να αυξάνονται αν υπάρχουν τέτοια συστήματα με τεράστιες και μεμονωμένες τράπεζες δεδομένων. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν έχετε δε ερωτήσεις με τα χαράς να απαντήσω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την προκλητική ε, επισκόπηση αλλά αυτό είχαμε ζητήσει ε, για να μπορούμε ε, να δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία την κατάσταση και το θέμα της πρόληψης πρέπει να μας απασχολήσει διαφορετικά και όπως άλλωστε και τις ευθύνες των εταιριών οι οποίες εμπλέκονται στο μέλλον μέλλον όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να προσάγεται στο δικαστήριο ο κλέφτης και όχι αυτός ο οποίος μας πούλησε ε, το ε, θησαυροφυλάκιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να ε, δικάσουμε τον κλέφτη και όχι ε, ε, συμφωνώ, αλλά εάν ο, ο τραπεζίτης τουλάχιστον πετάει τα λεφτά στην, ε, στο δρόμο θα πρέπει και αυτός να έχει κάποια συν, συνυπευθυνότητα για την κλοπή η οποία συνέβη στην τραπεζά του. Συμφωνώ. Έχετε ερωτήσεις από πλευράς των Ευρωβουλευτών. Ο Κρίστιαν. Ε, γερμανικά. Θα ήθελα να επανέλθω εις ε, το, ο, ε, στη βασική προϋπόθεση την οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα λέει ο κύριος Έλλερ διότι ε, υπάρχουν δύο ε, οπτικές γωνίες. Το ένα ε, σε σχέση με τη βιομηχανία του λογισμικού που πρέπει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των υπολογιστών και ξέρω ότι υπάρχει παραδείγματος χάρη εις την περιφέρειά μου ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων το οποίο δεν προστατεύεται και δεν είναι δυνατόν ε, να, ε, ε, να δαπανούμε εκατομμύρια για το cyberboard και να μην υπάρχει καμία προστασία. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το άλλο θέμα, δηλαδή μήπως υπερβάλλουμε όσον αφορά τις ρυθμίσεις και την προσπάθεια να ελέγξουμε τα πάντα. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα ε, σχετικά με την ασφάλεια. Αντιλαμβάνομαι ότι Υπάρχει το μήνυμα ε, ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό δεν είναι να αυξήσουμε την προστασία αλλά να μας απασχολήσει το ερώτημα εάν χρειαζόμαστε όλα αυτά, αν δεν πρέπει ίσως να τα μειώσουμε ε, και εάν δεν πρέπει να υπάρξει μία μειωμένη ε, μία μείωση των περιπλοκών των προγραμμάτων. Το άλλο όμως που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ε, εάν ε, η cyber security ε, φτάνει στα όρια μίας κοινωνίας η οποία είναι συνδεδεμένη μέσω του διαδικτύου υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταγωνισμός ε, από τη μία πλευρά από τις βιομηχανίες ε, να ανταποκριθούν ή στην κοινωνία που θέλει να είναι όλο και πιο στενά συνδεδεμένη και από την άλλη πλευρά της ασφαλείας που πρέπει να υπερισχύει. Σε ορισμένα λοιπόν συστήματα λογισμικού θα πρέπει να ε, υπάρχουν προγράμματα ε, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ δαπανηρά και το 50% των συσκευών στις οποίες ε, χρησιμοποιούνται δεν πρόκειται ποτέ να τα εκμεταλλευτούν. Επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό πρόβλημα τι είναι αυτό που μας απασχολεί, να έχουμε περισσότερη ασφάλεια ή εάν ή να θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια περιορίζει την δικτύωση της κοινωνίας αλλά χωρίς περισσότερη ασφάλεια λέει ο κύριος ε, Βάλτερ θα ήταν ε, ε, αμέλεια να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη διασύνδεση. Βέβαια η περιπλοκότηση είναι εχθρός της ασφαλείας. Όσο πιο περίπλοκα είναι τα συστήματά μας αυτομάτως τόσο πιο ανασφαλή γίνονται. Γι' αυτό και όταν είναι σημαντική η ασφάλεια και όταν πρέπει κανείς να βασιστεί εκεί πρέπει να έχει απλά προγράμματα και όσον αφορά την ε, ρύθμιση ή την υπερβολική παρακολούθηση στη δεκαετία του 60 και του 70 όταν ε, είχαμε ε, αρχίσει να χρησιμοποιούμε ίσως ζώνες θεωρούσαν στα αυτοκίνητα θεωρούσαν ότι ήταν κάτι περιττό. Εν όμως νομίζω ότι σώσανε πολλές ζωές εις ε, τις ε, οδικές μεταφορές και τώρα κανείς δεν ενοχλείται ότι πρέπει να φοράει ζώνη. Οπότε δεν πρέπει να απαιτήσουμε τα περίπλοκα συστήματα ε, να λειτουργούν όπως απαιτεί κανείς. Ας περιοριστούμε στα απλά. Επίσης, εάν χρησιμοποιούμε το Windows XP ε, θα, ε, ε, νομίζω ότι δεν αξίζει να χρησιμοποιήσουμε το πιο περίπλοκο πρόγραμμα ασφαλείας που υπάρχει γιατί και πόρους θα εξοικονομήσουμε και δεν θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια με αυτό. Σαφώς συμφωνώ με μερικά από αυτά που είπατε και διαφωνώ με άλλα. Ευτυχώς είμαι ο μόνος εδώ που δουλεύει για μια εταιρεία software. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που αφορούν αυτό το τομέα. Η απλοποίηση είναι κάτι καλό από απόψεως ασφαλείας. Μάλιστα, απολύτως. Όσο πιο πολύπλοκο είναι κάποιο λογισμικό, τόσο δυσκολότερο είναι να προστατευτεί Πόσο εύκολο είναι όμως να το προστατέψει κανείς. Χιλιάδες σελίδων γράφονται και τυπώνονται. Έχουν δημιουργηθεί ειδικέ οργανώσεις για να μειωθούν τα αδύνατα σημεία ενός προγράμματος, πώς θα μετεκπαιδευτεί το προσωπικό της χρήσης του, γενικά πώς χρησιμοποιείται αυτό το software πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλώς. Βέβαια δεν είναι ακόμη τέλεια η δημιουργία software και πάντοτε θα υπάρχουν τομείς που, όπου μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Και ακόμη και αν κάποιος γράψει ένα τέλειο λογισμικό, πάλι το λογισμικό αυτό, λόγω της χρήσης του, μπορεί να βλαφτεί, να δημιουργήσει μια λόγω ανθρω... λανθασμένης χρήσης. Είναι εύκολο λοιπόν να λέμε κάντε καλύτερο software και θα λυθούν όλα. Δεν ισχύει αυτό. Ακόμη και αν σας δώσω το καλύτερο δυνατό λογισμικό ασφαλείας μπορεί να τύχει κακής χρήσης ή να ξεχάσει κανείς να το ενημερώσει ή να το ανάψει καν και έτσι δεν θα προστατεύει. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα των αυτοκινήτων. Εδώ Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, δεν ισχύει απόλυτα. Γιατί, διότι ένα αυτοκίνητο, οποιοδήποτε, ε, δημιουργείται, στα, ε, λειτουργεί στατικά, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μισή Φεράρι και μισό ΦΙΑΤ μαζί. Επίσης όταν το οδηγούμε στο δρόμο δεν υποτίθεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά αν συνεχώς του επιτίθενται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον υπολογιστή. Τον αλλάζουμε συνεχώς και πολλές φορές υφίσταται επιθέσεις κάθε φορά που μπαίνει online. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να προστατευτεί ο υπολογιστής. Για να αναφερθώ τώρα σε αυτό που είπατε για το online και το offline ως προς την ασφάλεια. Εδώ βλέπουμε online με έναν αντικατοπτρισμό αυτού που συμβαίνει offline δηλαδή. Μπορεί να θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος θέλει περισσότερη τεχνολογία και θα τη χρησιμοποιήσει ούτως ή άλλως ίσως και λάθος, ίσως και άσκημα, ίσως γιατί δεν την καταλαβαίνει καλά ή δεν ξέρει ποιοι είναι οι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια. Και γι' αυτό το θέμα είναι να δημιουργηθούν ήθη ασφαλείας, ασφαλιτικά ήθη. Ιδιαίτερα αν δεχτούμε αυτά που ακούστηκαν πριν, ότι είναι και ευθύνη, είναι ευθύνη και του χρήστη η ασφάλεια. Αν δεν μάθει ο χρήστης ποια είναι η σωστή χρήση, δεν θα κάνει τη σωστή. Και εγώ θα ήθελα να επανέλθω ε, στο εάν υπάρχει ένα ασφαλές ε, σύστημα το οποίο καλύπτει 4 ε, εκατομμύρια άτομα στην Γερμανία. Δεν πιστεύω ότι είναι ασφαλές το σύστημα αυτό και ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα διαφορετικά για να αποφύγουμε ε, τα ε, γεγονότα που ε, συνέβησαν στην Ελβετία τελευταίως. Ε, υπάρχει όμως ε, ε, το γεγονός ότι αν μία εταιρεία είναι επιτυχής θα τις επιτεθούν και κάποια στιγμή θα πετύχουν. Αλλά έτσι δεν μπορούμε να δικτυωθούμε περισσότερο. Υπάρχει το σύστημα ασφαλείας Καπέρσκι παραδείγματος χάρη. Μπορούμε ίσως να έχουμε συστήματα τα οποία δεν θα είναι είναι για τα κρατικά μυστικά, αλλά πρέπει να δούμε τι χρειάζεται ο απλός χρήστης, ο οποίος δεν μας ζητά, δεν απευθυντούνται σε Μάντεκ ούτε στις δικές μας εταιρείες. Θέλουμε μεν να αυξηθεί η ασφάλεια, να, τώρα αρχίζουν να υπάρχουν πιο ασφαλή ε, λογισμικά αλλά τι θέλουμε θέλουμε να είναι ε, απολύτως ασφαλή ή θέλουμε να έχουμε συστήματα που θα είναι εύχριστα στο μέλλον ε, θα δώσω τον λόγο εις τους μιλητέ, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τμήμα αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι εδώ αναφερόμαστε μόνο στις αμερικανικές εταιρείες και στους Αμερικανούς και στους Κινέζους δηλαδή ε, όποιος θέλει να έχει καταναλωτές και να τους προσελκύσει θα πρέπει να ε, τους εξυπηρετεί και πρέπει να δούμε και εμείς πολιτική εάν μπορούμε να βοηθήσουμε ένα προϊόν με το να βελτιώνουμε το λογισμικό και να το καθιστούμε πιο ασφαλές. Και με αυτό το ερώτημα θα σταματήσω εδώ διότι νομίζω ότι το ποινικό δίκαιο είναι ο τελευταίος, το τελευταίο τελευταίο για να προβούμε σε κυρώσεις αλλά ακόμη και αν κανείς δεν ε, ε, πεθαίνει υπάρχουν πολύ σημαντικές οικονομικές βλάβες και ζημίες που μπορούν να προκληθούν και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς εμείς στα πλαίσια της εργασίας μας σαν Ευρωβουλευτές μπορούμε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά και θέλω τώρα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και να παρακαλέσω τους ομιλητές για το τρίτο και το τέταρτο μέρος να έρθουν. Ε, θα πάρουμε τις δύο ενότητες μαζί κατά τρόπον ώστε ε, στη συνέχεια να έχουμε μία ώρα ερωτήσεων για τα έξι τμήματα, τέσσερα τμήματα και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα μαζί. So, um, Κυρίες και κύριοι, τρίτος και τέταρτος γύρος. Να σας κάνω όμως και μια εισήγηση. Το Κοινοβούλιο ευχαριστεί τους αδέλφους της Επιτροπής Λίμπε και η τρεκέ βιομηχανίας γιατί η Λισαβόνα άλλαξε τη στάση του Κοινοβουλίου ως προς το πώς θα έπρεπε να εφαρμόζει τα νομοθετικά του καθήκοντα. Στο Κοινοβούλιο μέχρι τώρα βασίλευαν οι εισηγητές και οι εισηγήτριες. Αυτό αλλάζει και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί κυρία Χολμάγερ είχε τόσο συνεργατική στάση για την εξέταση αυτού του θέματος και οι συνάδελφοι από την Ήτρε το εξετίμησαν αυτό δεόντως γιατί όλα σχετίζονται τα θέματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κατά πόσον πρέπει η ενίσα να έχει παρατεταμένη εντολή ή όχι. Και έτσι ερχόμαστε σε ένα σημαντικό ερώτημα που θα είναι το θέμα του τρίτου γύρου, η συνεργασία μεταξύ οργάνων. Όταν άρχισα την κοινοβουλευτική μου θητεία, ήμουν και εγώ εισηγητής πριν από πολλά χρόνια και οι μεγάλες για να το πω έτσι χώρες μέλη δεν ήθελαν να δημιουργηθεί το ΕΝΙΣΑ γιατί έλεγαν ότι είναι εθνικό καθήκον και ιδιοδοσία. Η κυβερνοασφάλεια. Δεν θεωρούσαν ότι μπορούσε ή έπρεπε η Ευρώπη να παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό το θέμα. Η στάση αυτή άλλαξε και τώρα θεωρούμε ότι χρειάζεται, έχει ένα καθήκον και το ενωσιακό επίπεδο ας πούμε τις διαπραγματεύσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς διαδρούν δηλαδή οι χώρες μεταξύ τους ας πούμε. Θεωρήσαμε λοιπόν σημαντικό εν ώψη του επικρεμαμένου νομοθετήματος να δούμε πρώτα ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι προϋποθέσεις αυτής της διαθεσμικής συνεργασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε εδώ εκπροσώπους με νομική μορφωσή τον κύριο Αμπάση που θα είναι ο αντιπρόεδρος του γύρου η δόκτωρ Βικτόρια Μπέινς από την Ευρωάστα, πρόσωπος της ΕΝΙΣΑ και θα αρχίσουμε με το ΕΝΙΣΑ. Συμφωνείτε και εσείς, συμφωνείτε. Και αρχίζω ερωτών. Τι εννοείται συνεργασία, ποιες είναι οι ελλείψεις της γιατί στα πλαίσια του ορίζοντος του 2020 κανένα μέλος της ΕΝΙΣΑ δεν παρακάθισε εδώ να μας συμβουλέψει παρά το ότι επρόκειτο για 250 εκατομμύρια Εγώ έχω συνεργαστεί με το Αμερικανικό ΝΙΣΤ αλλά δεν ήρθαν και τότε να μας δουν ούτε το ΕΝΙΣΑ ούτε άλλες γενικές διευθύνσεις. Επομένως υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα οριζόντια συνεννόησης και στην Κομισιόν και μεταξύ άλλων οργάνων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποιο επίπεδο συνεργασίας απαιτείται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν από απόψεως ενίσας να μας πούν τι καλό ή τι κακό παράδειγμα υπάρχει, τι βελτίωση μπορεί να γίνει. Ορίστε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να με εκπροσωπήσω την Ενίση εδώ σήμερα. Να ξεκινήσω μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ε, παλιάς και της ασφάλειας των πληροφοριών, αυτό που κάνουμε τα 15-20 χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν αναμένω μια απάντηση. Να σας πω ότι πιστεύουμε εμείς. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι θέμα προοπτικής. Όταν μιλάμε για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εξετάζουμε το θέμα τη. Ασφάλιση των πληροφοριών σε, από μια διεθνή σκοπιά, δηλαδή δεν ε, θα αναφέρεται κάποιος σε έναν αξιωματικό ε, για την ασφάλιση στον κυβερνοχώρου σε μια μικρή επιχείρηση, αλλά το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρου έχει να κάνει με τη συνεργασία. Σήμερα θέλω να σας πω ότι με αυτό ασχολείται και η ενίσχυση, ενδυνάμωση. Ε, μάλλον η δύναμη της ενίσα ε, και η κύρια αποστολή της είναι να προωθήσει ένα ισχυρό πολιτισμό ασφάλειας των πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν σήμερα για, σε αυτό θα μιλή, για αυτό το θέμα θα μιλήσω, δεν θα αναφερθώ σε τεχνικές πτυχές και θα σας πω πώς προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το όραμα. Ας ε, ξεκινήσουμε ε, με παρουσίαση του οργανισμού είμαστε 16 ε, άτομα και πρέπει να εργαζόμαστε σε συγκεκριμένο τρόπο και δημιουργηθήκαμε το 2004. Έχουμε ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνη, το αποκαλούμε κέντρο εμπειρογνωμοσύνη. Ελπίζω να με θεωρείτε ότι υπερηφανευόμαστε. Έχουμε κάποιες, ε, κάποιους εμπειρογνώμονες στην υπηρεσία, αλλά θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά εργαζόμαστε μέσω μόχλευσης της εμπειρογνωμοσύνης στα κράτη-μέλη, δηλαδή συστήνονται ομάδες και χρησιμοποιούμε και πυρογνώμονες στα κράτη-μέλη για να επιλύσουμε διασυνοριακά προβλήματα. Υποστηρίζουμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ε, σε όλο το θέμα των ε, πληροφοριών πληροφορικής και ανταλλάσσουμε πληροφορίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν, ας περάσουμε στην εργασία με τα κράτη-μέλη. Ε, Ένα πολύ σημαντικό στόχο τη ΕΝΗΣΑ είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή εμπειριών και βελτιστών πρακτικών μεταξύ των κρατών μέλων. Εμεί προσθέτουμε τι δικέ μα ιδέε και όσα έχουμε μάθει από τα διάφορα project στην εξίσωση, αλλά τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή των πρακτικών και διδαγμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό και με τη διαμεσολάβηση μεταξύ των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών οικοδομούμε μια ευρεία προσέγγιση. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή στα 60 άτομα, αλλά εργαζόμαστε με όλου του εμπειρογνώμονε εκεί, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, η Ενίσα ε, το 2008 ήταν ένας οργανισμός ε, activity based, ε, βασιζόταν σε δραστηριότητες, δηλαδή ας κάνουμε κάτι για τις υποδομές, ζωτικής σημασίας, κατόπιν γίναμε ένας οργανισμός που επικεντρώνονταν στα αποτελέσματα, ενώ τώρα ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε τον αντίκτυπο. Έχουμε μόχλευση της ε, εμπειρίας ε, στην αγορά. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την παρουσία μας στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει το πρόβλημα, να είμαστε σίγουροι ότι ασχολούμαστε με τα πρακτικά προβλήματα που συναντούν τα κράτη-μέλη σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν θέλουμε να βγάλουμε τους ανθρώπους εκεί, ε, να υπάρχει κινητικότητα και να υπάρχει ευρία κάλυψη. Εδώ βλέπετε πόσα πολλά κάνουμε. Συνεχώς ταξιδεύουμε σε τις χώρες ε, και συζητούμε με ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. αυτό είναι ο πυρήνας των εργασιών μας. Επίσης, συνεργαζόμαστε και με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλους φορείς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει προσθεμένη αξία στη δράση της ΕΝΗΣΑ, δηλαδή δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτά που κάνει η Κομισιόν ή άλλα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμοί. Ξοδεύουμε πολύ χρόνο να ευθυγραμμίζουμε τις πρακτικές μας και τους στόχους μα. με Άλλου ευρωπαϊκού φορεί και όργανα. Σα έχω δώσει ορισμένα παραδείγματα. Συνεργαζόμαστε με την κόμμα, με τη γάμα Δέλτα Ίφσο, τη γάμα Δέλτα Enterprise, συνεργαζόμαστε με το JRC, το Ερευνητικό Κέντρο, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, υποστηρίζουμε το νέο θεσμικό υπάρχει μνημόνιο συνεννόηση με το ETSI και ε, προετοιμάζουμε ένα με τη ΣΕΝ και έχουμε ε, καθεστώς παρατηρητή στην ομάδα εργασίας ISO ε, CS27 και έχουμε και μόνο κατανόησης με την Ευρωπόλ. Τώρα, ο ιδιωτικό τομέα πάρα πολύ σημαντικός γιατί ε, οι περισσότερε υποδομέ ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε δηλαδή ευρείε επαφέ με τον ιδιωτικό τομέα και διαθέτουμε αυτό το δίκτυο στα κράτη-μέλη. Συναντούμε συχνά ε, άτομα από τη βιομηχανία. Για να σας πω ένα παράδειγμα, ευρωπαϊκό ΣΔΙΤ για την ανθεκτικότητα, ε, στο οποίο ακούσατε μια-δυο φορές σε αυτήν την ακρόση και η εκπρόσωποι του Διευθυντικού τομέα συμμετέχουν στα περισσότερα από τα project μας. Ε, κύρια μηνύματα, πώς φέρνουμε τις κοινότητες κοντά. Μπορεί να είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα να φέρουμε κοντά τις κοινότητες παρά τα κράτη-μέλη, γιατί υπήρχαν αρκετά μεγάλα εμπόδια ανταλλαγής προφοριών μεταξύ των κοινοτήτων Λοιπόν, Τώρα έχουμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα που ανοίγει τι πόρτε σε μεγαλύτερο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών αυτών, αλλά πρέπει να διανύσουμε μακρύ δρόμο. Σε ορισμένε περιπτώσει ξέρουμε ότι κάνουμε τα ίδια με ε, σε τέτοια εγχειρήματα που έγιναν από άλλου, κοινότητε άλλες ε, stakeholders και δεν ανταλλάσσουν πληροφορίε. Αυτό είναι κάπως τρελό και φυσικά δεν συμφέρει οικονομικά. Δεν έχω πολύ χρόνο. Θα σας αναφέρω την πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση, ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι κάνει η ΕΝΙΣΑ. Ε, αυτό ε, προέκυψε από το σχέδιο δράσης της Κομισιόν του 2009 ε, η προθεσμία του 10.000 προήρθε από την ε, Υπουργική. Πολύ χώρα στη συνέχεια. Είχαμε μικρό αριθμό κρατών μελών, όμως ε, είχαμε τελικά 27 κρατημέλη μέλη στην χώρες της ΕΖΕΣ. Μεγάλο παράδειγμα, δηλαδή πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι μικρό και να καταλήξουμε σε κάτι που συμμετέχουν όλοι. Τι δοκιμάσαμε. Κάποια πολύ απλά πράγματα και ακόμη και αν ελέγξαμε αυτά τα πράγματα. δεν ήμασταν τόσο καλοί, βέβαια βελτιωνόμαστε. Δοκιμάσαμε αν δεχτεί επίθεση ένα κράτος μέλος, από ένα κράτος μέλος παραδείγματος χάρη, ποιον θα πάρει τηλέφωνο δεν είναι τόσο προφανέ ήδη αυτό. Ακόμη λιγότερο προφανές είναι πόσο καλή είναι η κατανόηση τη εξουσία αυτού του ανθρώπου να λαμβάνει αποφάσεις και τις εντολής του. Αυτό είναι ζωτικό. Δεν θα σε περάσει μισή ώρα μιλώντα με κάποιον που δεν μπορεί να σε βοηθήσει τελικά. Και επίση ε, τι, τι χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία. Όπως είπα, συμμετείχαν όλα τα κρατημέλη τη χώρες τη ΕΖΕ, στο προφίλ, συμμετείχαν ήταν Υπουργοί, Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, κοινότητες EAP και άλλοι σχετικοί stakeholders, 70 οργανώσει και 150 εμπειρογνώμονε και νομίζω ότι η γενική εντύπωση είναι ότι άξιζε αυτό το εγχείρημα και ήταν ένα καλό βήμα προς ε, ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο ε, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ε, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα να δοκιμάσουμε έτσι λοιπόν. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε συγχωρείτε αυτές τις ασκήσεις για να δημιουργήσουν κάποιους θύλακες πολιτικής, για να έχουμε ένα διασυνοριακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να σας πω ε, τα πορίσματα διατίθενται και στην ιστοσελίδα μας. Φυσικά όλα είναι δωρεάν, πηγαίνετε να το επισκεφτείτε. Πολύ ενδιαφέρον το υλικό για όλες τις ομάδες stakeholders και για τον ιδιωτικό τομέα. Τα πορίσματα είναι οικοδόμηση εμπιστοσύνη, σχεδιασμό και δομή, συνεννόηση, σημεία επαφή και όπω σα είπα θα έχετε πλήρη κατάλογο συστάσεων. Τώρα, ετοιμαζόμαστε για την πρώτη κοινή άσκηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, που ε, ανακοινώθηκε από τις Κρούς και Ναπολιτάνο στην ε, Ουγγαρία νωρίτερα φέτος. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Συμπεράσματα. Λοιπόν, τι θέλω να καταθέσω εδώ, ότι... Λοιπόν, κύριε κυρία τι τη διευκολύνει το διάλογο μεταξύ κρατών μελών, θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΕΝΑΙΕΣ. Φυσικά πρέπει να μα καλέσουν και ω ένα οργανισμό που έχει να κάνει με τι βολιστικέ πρακτικέ μπορούμε να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία να αντιμετωπίσει καθημερινές προκλήσεις σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Να σας πω ότι έχουμε και κάποια σχόλια επί της οδηγίας, αν έχω χρόνο. Πιστεύουμε ότι η οδηγία είναι ένα πολύ καλό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Σε ανταποκρίνεται στις περισσότερες ανάγκες μας, έχω κάποια σχόλια. Το πρώτο είναι να μην βλέπουμε στη τεχνολογία, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα ε, στο λογισμικό, έχουμε το virtualization, τις εφαρμογές, ε, πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε το ότι μπορεί να παρακολουθούμε τα δεδομένα σε πολλά επίπεδα και φυσικά αυτό αναμένουμε να κάνουν και οι αρμόδιοι. Συμφωνούμε με τις ποινές, θεωρούμε ότι είναι ανάλογες με τον δίκτυπο των κλίματος, όμως πρέπει να είστε προσεκτικοί με τις τεχνικές μέτρησης, Ο ρυθμός των bot στα botnets, παραδείγματος χάρη, του προγραμμάτων, δεν είναι καλό εργαλείο μέτρηση σε σχέση με τον αντίκτυπο. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν κάποιοι ορισμοί να βελτιωθούν, κυρίως ό,τι αφορά πρόσβαση, interception of data, δηλαδή υποκλοπή δεδομένων. Ε, νομίζω ότι καλό είναι να τα ξαναδείτε αυτά. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε δύο επίπεδο πρόσβαση και αποκλοπή δεδομένων μπορεί να εφαρμοστούν νομικά χωρί τη συγκατάθεση του, του κατόχου του συστήματο πληροφοριών, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την ε, ε, υποκλοπή, παραδείγματο χάρη, από του αστυνομικού ε, για να διαλύσουν τα botnets και στο ε, άρθρο 41 θεωρήσαμε ότι εκεί είναι κάπως αδύναμη η διάταξη και δεν υπάρχει προτυποποίηση ενώ θέλετε να υπάρχει διαπερίοδος ε, μεταξύ που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη και στο άρθρο 15 μπορεί να σκεφτείτε να βάλετε την Ενίσα και την Europol ε, ως ε, παραλήπτες των δεδομένων. Η Ενίσα ήδη λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 13α ε, της νομοθεσίας για τις λεπικοινωνίες, κάποιες κοινοποιήσεις για τις παραβιάσεις ε, απειλών. Μπορείτε να μας προσθέσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο επόμενος ομιλητής ε, προέρχεται από το Eurojust ε, από ό,τι ξέρω είστε επικεφαλής μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων που εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις και καλό θα ήταν να έχουμε μία καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, θα έπρεπε Ε, γι' αυτό το λόγο να ε, εξετάσουμε και αυτή την πτυχή για την νομοθετική πρόταση την οποία εξετάζουμε. ημέρα σας. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά όπως θα διαπιστώσετε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, και τον κύριο Μάγερ που με προσκάλεσε. διότι ε, βλέπετε εδώ έναν ε, νομικό ή με δικαστικός ε, πρώην εισαγγελέα και θα κοιτάξω τη δικαστική πτυχή. Αυτά που άκουσα είναι πολύ ενδιαφέροντα διότι είναι τόσο μακριά από αυτά τα οποία σκέφτονται οι δικαστικοί οι δικαστές και οι εισαγγελείς ε, ε, στο χώρο τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς εμείς αντιμετωπίζουμε ε, τις, τα κυβερνοεγκλήματα και τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε όπως το κέντρο της κυβερνοεγκληματικότητας. Ξέρω ότι όλοι γνωρίζετε τι είναι το Eurojust αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για έναν οργανισμό, για μία μονάδα δικαστικής συνεργασίας που υπάρχουν μόνο εισαγγελείς και δικαστές και όπου ασχολούμαστε με ε, ε, εγκλήματα και αξιόπινες πράξεις και στα πλαίσια της Eurojust έχουμε ε, οργανώσει έχουμε οργανωθεί με διάφορες ομάδες σκέψεως και ομάδες εργασίας ακριβώς για να τονίσουμε ορισμένες δικαστικές ψυχές που είναι πολύ περίπλοκες. Υπάρχει λοιπόν ε, ε, υπάρχει η μονάδα της, ε, των οικονομικών εγκλημάτων την οποία προεδρεύω και έχει σαν στόχο τον, την καταπολέμηση της της ε, εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Οι ε, υπεύθυνοι λοιπόν που είναι σε αυτό το χώρο, οι περισσότεροι, είναι ειδικευμένοι και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, διότι αντιλαμβανόμαστε στην Eurojust και στις ανταλλαγές που έχουμε με τους δικαστικούς, έχουμε και την ε, Europol που υπάρχουν τεχνικοί, αλλά οι οι δικαστές δεν είναι καθόλου ειδικευμένοι σε αυτό το χώρο. Οπότε ε, στην ε, ε, ομάδα αυτή της Eurojust υπάρχουν οικονομολόγοι και οι δικαστικοί οι οποίοι προσπαθούν να συνεργαστούν και να δούμε μεταξύ τεχνικών και δικαστικών πώς μπορούμε να εξαρθρώσουμε τέτοια δίκτυα εγκληματικά. Έχουμε ένα δημόσιο χώρο στο διαδίκτυο στη Γαλλία, τον οποίο, ο οποίος υπέστη μία επίθεση και επί μέρες ε, δεν μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση. Όταν ε, μας ενημέρωσα στην Eurojust, εγώ ήθελα να λύσω το πρόβλημα στα πλαίσια αυτής της ομάδας, γιατί ο Γάλλος ε, δικαστής προσέφυγε βάσει του τι έκανε η αστυνομία χωρίς να γνωρίζει τις τεχνικές ιδιομορφίες. Άκουσα ιδίω ε, τον εκπρόσωπο της εταιρείας Χάος ο οποίος ε, εξηγούσε πώς ε, καταλήξαμε σε μια κατάσταση όπου μπορούν να ευθύνονται οι υπεύθυνοι των τραπεζών αλλά πριν προσδιορίσουμε αυτή την συνυπευθυνότητα πρέπει να ξέρουμε γιατί ομιλούν οι δικαστικοί και τι ε, κάνουν. Πρέπει δηλαδή να δούμε ε, την ε, περίπτωση αυτή μιας επιθέσεως σε μία ιστοσελίδα να δούμε πώς, μπορούσαμε, πώς μπόρεσαν από δύο ανατολικές χώρες εκ των οποίων μία ήταν η Ρουσική Ομοσπονδία να υπάρξει μία επίθεση σε μία ιστοσελίδα στη Γαλλία δηλαδή μία ολόκληρη ενημέρωση η οποία μπορεί να ήταν χαμιανός χρόνος αλλά ήταν ενημέρωση των δικαστικών για να καταλάβουν το θέμα. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να βοηθήσουμε τους δικαστές και τους δικαστικούς στο, στην αντιμετώπιση αυτών των αξιοπίνων πράξεων ε, και τώρα γιατί αξιόπινες πράξεις μιλάμε. Ε, προηγουμένως ε, ελέγχθη ότι υπάρχουν διάφοροι κατάλογοι των αξιοπίνων ε, πράξεων στο ε, διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο και θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινό ορισμός και αυτό είναι σωστό διότι μεταξύ των διαφόρων χωρών δεν συμφωνούν οι ε, εθνικοί εκπρόσωποι για το τι θεωρούν μία επίθεση στον κυβερνοχώρο και εφόσον δεν συμφωνούν δεν μπορούν να συντονιστούν και με, όλες με όλα τα επακόλουθα δηλαδή να ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος ε, σε ποια ε, νομοθεσία, ε, για ποια αξιόπινη πράξη πρόκειται, τι παραγραφή υπάρχει, αν είναι αξιόπινη πράξη, αν είναι απλώς αδίκημα, παράπτωμα ή ποινικό, ποινικό αδίκημα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι ορισμοί τους οποίους πρέπει να καθορίσουμε και θα σας σας πω ε, πώς εμείς ε, εξετάζουμε τους ορισμούς της οδηγίας στο άρθρο 34. Καταρχήν να σας πω ότι στην Eurojust πέρυσι το 2010 ανοίξαμε 32 φακέλους για ε, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και τώρα βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο φακέλων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν μόνο 32 περιπτώσεις στα 27 κράτη-μέλη, δηλαδή μόνο 32 υποθέσεις για έναν ολόκληρο χρόνο. Πρέπει λοιπόν και θα επανέλθω στο σημείο αυτό να δείξουμε και να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν να συντονιστούμε στα πλαίσια αυτά. Γιατί σας λέω μόνο 32 υποθέσεις το 2010 ε, ενδέχεται φέτος κάπως να αυξηθούν αυτές οι στατιστικές. Ήθελα όμως να σας πω ότι η υπεύθυνοι της ε, καταπολέμησης ε, της κυβερνοεγκληματικότητας είναι σε τρία επίπεδα καταρχήν η δικαστική και η αστυνόμη δεύτερον οι αρχές όπως το Eurojust και το Europol που συνεργάζονται τρίτον τρίτο επίπεδο και αυτό θα το θίξουμε ε, συντομία μετά εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως Δηλαδή μπορεί να συνεργαζόμαστε, μπορούμε να προχωρούμε από κοινού, αλλά άπαξ και συνεργαστείτε με άλλες χώρες είμαστε υποχρεωμένοι να βασιστούμε ε, σε διεθνή νομικά εργαλεία. Αναφέραμε την συνθήκη της Βουδαπέστης. Ελάχιστα κράτη όμως έχουν κυρώσει αυτή τη συνθήκη. Άπαξ λοιπόν και βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν υπάρχει μία ε, δικαστική πλειοψηφία για να συνεργαστούμε. Στην περίπτωση που σας ανέφερα προηγουμένως στη Γαλλία ε, βρίσκουμε ότι η υπεύθυνη είναι στη Ρωσία και με ε, συνεργασίες ε, δυσκολευόμαστε πολύ για να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία. Ε, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια του, της Eurojust και στην επιθυμία να λύσουμε αυτές τις αξιόπινες ε, πράξεις. Πρώτον, ενημέρωση. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση των ε, νομικών. Ε, δεύτερον, ανταλλαγή πληροφοριών. Το προβλέπει η οδηγία. Ναι, ε, εδώ προβλέπεται ότι πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και αναφέρεται στα σημεία επαφών. Εφιστώ την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν ήδη ορισμένα σημεία επαφής και το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει ε, αυτά τα ίδια σημεία να ισχύσουν και στο μέλλον. Και είναι πολύ βασικό να επιμείνουμε σε αυτά τα σημεία επαφής, διότι πολλές φορές η ε, ε, ε, δικαιοδοσία ε, στη μία χώρα ή στην άλλη θα πρέπει να έρθει σε επαφή με αυτά τα σημεία επαφής για να μπορέσει να αποκομίσει πληροφορίες. Και δύο τελευταίες δυσκολίες. Η πρώτη αναφέρεται στην ταχύτητα ε, αυτών των αξιοπίνων πράξεων που απαιτεί άμεση αντίδραση και ε, πρέπει να προβλέψουμε κανόνες πιο ευέλικτους ε, σχετικά με τη δικαιοδοσία ε, και υπάρχει και το πρόβλημα των τρίτων κρατών που προανέφερα. Καταλήγοντας λοιπόν, θεωρώ ότι η οδηγία όπως παρουσιάζεται είναι αρκετά καλή γιατί είναι αρκετά γενική, σφαιρική, διότι είναι οδηγία όχι κανονισμός. Πρέπει να ενισχυθεί σε ορισμένα θέματα για τα σημεία επαφής ε, τον καθορισμό των ατόμων που θα είναι αποτελεσματικά και χρήσιμα, την ε, συμμετοχή των τρίτων χωρών και τη δημιουργία ενός κέντρου ε, ε, ε, εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταρτήσει μία ομάδα που προσπαθεί να προωθήσει αυτό το κέντρο και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει μία καλύτερη τεκμηρίωση και κατάρτιση των δικαστικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και... Ευχαριστώ σας, είμαι και εγώ πάρα πολύ ευγνώμων. Ε, νομίζω ότι η ιδέα της κυρίας ε, Χολμάιερ να εμπλέξει την Eurojust διότι από πλευράς ε, των εθνικών εισαγγελιών πρέπει, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και των θεμάτων τα οποία θεωρούνται αξιόπινα στα διάφορα κράτη-μέλη. Για να προχωρήσουμε όμως τώρα στην επόμενη ομιλία κυρίου Μπέιν της ε, Europol, της, της κυρίας Μπέινς της Europol αντιλαμβάνομαι ότι ε, και εσείς ε, έχετε κάποια συνεργασία με τους Ευρωπαίους πολίτες κατά τρόπον ώστε να ενημερώσετε για την διάσταση αυτής της εγκληματικότητας των κυβερνοχώρων για να υπάρξουν ορισμοί και το άλλο θέμα θέμα βέβαια είναι ε, τι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα ο Ευρωπαίος πολίτης εάν ε, γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και εάν ε, πλήτεται από την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και την οπτική γωνία της Europol και καλό θα ήταν να συζητήσουμε το θέμα αυτό και σας δίνω το λόγο. Thank you very much. Good afternoon, ladies and... Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΕΛΕΦ και την κυρία Χόλμαγερ γιατί προσκάλεσε την Ευρωάστ σήμερα. Η θέση μας και εδώ και για προς στην πρόταση είναι νομίζουμε ιδιαίτερα επίκαιρες γιατί αυξάνονται οι επιθέσεις κατά πληροφορικών συστημάτων και οι κυβερνοεπιθέσεις γενικότερα. Αλλά ιδιαίτερα εκτιμούμε τη συνεργασία που εκτιμάται όλο και περισσότερο στην Ένωση μεταξύ ελληνικών οργάνων. Για όσους δεν γνωρίζετε καλά την Ευρωάστ, είμαστε το κυριότερο κέντρο της Ένωσης για τεχνογνωσία ως προς την επιβολή του νόμου. Μεταξύ των υπηρεσιών μας Έχουμε ειδικού για έρευνες σε χώρες μέλη, για σήμανση, για συνδυασμό για συνδυασμένες έρευνες για διαμεθοριακά προβλήματα και δίνουμε στρατηγικές κατευθύνσεις. Επίσης υπηρετούμε σαν κέντρο πληροφοριών για τα εγκλήματα στην Ευρώπη, ταυτίζουμε ο, στοχευμένες ομάδες και δίνουμε πληροφορίες με βάση τους φακέλους που διαθέτουμε, τους αναλυτικούς φακέλους που διαθέτουμε. Εκτός αυτού έχουμε ένα on-site δίκτυο 140 αξιωματούχων από διοκτικές αρχές στην Ένωση και τρίτες χώρες και άλλους ειδικού για τα κυβερνοεγκλήματα, ιδιαίτερα από το Serious Organized Crime Agency του Ηνωμένου Βασιλείου και την FBI. Πέρυσι η Ευρωάς δημοσίευσε μία αξιολόγηση του κινδύνου για το έγκλημα στο ίντερνετ λεγόμενο η όκτα. Αυτή η μελέτη έδειξε τι ρόλο παίζουν τα botnets και επίσης έδειξε ότι διευκολύνουν την ε, μεγάλης κλίμακας, τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις σε πληροφορικά συστήματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διάλυσή τους είναι προτεραιότητα. Αναγνωρίζοντας ότι τα ίδια κυβερνοεγκληματικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και έχοντας παρατηρήσει ότι οι διαχωρισμοί μεταξύ διαφόρων τύπων ίντερνετο εγκλημάτων ταυτίζονται όλο και περισσότερο και οι χώρες μέλη και οι οργανώσεις της Ένωσης άρχισαν να συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν το κυβερνητικό έγκλημα. Η ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι επίση υψηλή προτεραιότητα, αλλά επίσης και η δημιουργία στενότερης συνεργασίας με άλλες ε, ενωσιακέ υπηρεσίες. Θα σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας για τη δικαστική συνεργασία η Ευρωπόλ και η Ευρωδίκ φυσικά συνεργάζονται πολύ στενά. Η Ευρωδίκ είναι μέλος όχι μόνο του ανάλυσης Workfile Cyborg αλλά και μέλος της ε, ομάδας Task Force για το κυβερνοέγκλημα της Ευρωένωσης που χρηματοδοτείται από την Ευρωάστ οι δύο υπηρεσίες συνεργάζονται άμεσα για στρατηγικά και λειτουργικά θέματα και τα περισσότερα παραδείγματα αφορούν περιπτώσεις που ακόμη ερευνώνται. Ορίστε ορισμένα παραδείγματα από τον ευρύτερο κυβερνοεγκληματικό χώρο. Πρώτον υπάρχει μια έρευνα που συνδυάζει που οργανώνει η Ευρωδίκ με χρηματοδότηση από το EU Emissions Trading System και που έχει καταφέρει να ταυτίσει <clears throat> τις χρηματοδοτικές ροές και να πληροφορήσει τις χώρες μέλη για την εγκληματική συμπεριφορά των ενδιαφερομένων ομάδων. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει ένα σχέδιο βάσει του οποίου τα χρήματα που προέρχονται από το κυβερνοέγκλημα ξεπλένονται. Και εδώ η ανάλυση της Ευρωάστα βοήθησε τους εισαγγελείς και άλλους διώκτες να κάνουν αποτελεσματικότερη διαμεθοριακή έρευνα. Η συνεργασία μας με την Ενίσα είναι πιο πρόσφατη αλλά το ίδιο σημαντική. Τη στιγμή που μιλάμε η Ενίσα και η Ευρωάστα συνοργανώνουν ένα ε, εργοαστήριο στην Πράγα για να δημιουργήσουν στενότερες σχέσεις μεταξύ χωρών μελών, διοικητικών αρχών των χωρών μελών και ομάδων ε, ανταπόκρισης ηλεκτρονικά. Οι μεν ε, διερευνούν εγκλήματα, οι δε έχουν, δίνουν, θέλουν να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές και αυτά είναι συμπληρωματικές δραστηριότητες και καταλήγουν σε κοινέ αναφορές και αναλύσεις για τις απειλές και τους κινδύνους. Η προτινόμενη λοιπόν δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κυβερνοεγκληματικού Κέντρου το 2013 είναι κάτι το επίκαιρο. Η Ευρωπόλ θέλει να παίξει ένα ρόλο στην συλλογή πληροφοριών και στις έρευνες του κέντρου αυτού και επίσης θεωρεί ωφέλιμο να συμμετάσχουν και ειδικοί από την Ευρωδίκη και την Ενίσα. Προβλέπεται παραδείγματο χάρη να υπάρξουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του κέντρου και του EU CERT, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ηλεκτρονικής Ανταπόκρισης. Εμείς λοιπόν δεχόμαστε την ποινικοποίηση της παραγωγής, πώληση, χρήσης, διάθεσης για χρήση, εισαγωγής κτλ. κυβερνοεγκληματικών εργαλείων. Επίσης, συμφωνούμε με την εφαρμογή μια συγκεκριμένης κατηγορίας που να επιτρέπει τη σύλληψη και την ε, μεγαλύτερη συνεργασία και ενδυνάμωση των, 20, ε, των ε, σημείων επαφής χωρίς διακοπή. Ως προς τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τις κυβερνοεπιθέσεις η Europol ταπεινά προτείνει να, δοθεί να γίνει περισσότερη ανάλυση του κατά πόσον θα αφορά όλες τις, αυτές τις επιθέσεις ή μόνο όσες θεωρούν τα κράτη-μέλη ως ιδιαίτερα σημαντικές. Εφόσον η πρόταση λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν τι αποτελεί σημαντική ζημία για αυτά, μπορεί να καταλήξουμε σε ασυνεπή συμπεράσματα που δεν θα επιτρέπουν αποτροπή. Και τέλος, προς πληροφόρησή σας, θα ήθελα να σας τονίσω ότι υπάρχει και ένα σχέδιο που αναλύεται αυτή τη στιγμή να απλοποιηθούν οι αναφορές κυβερνοεγκλημάτων από τα κράτη-μέλη στην Ευρωάστ. Είναι το σύστημα ICROS που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συλλέγονται τέτοιου είδους αναφορές και άρα να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ο νομοθέτης. Σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπέινς. Αυτή τη στιγμή βέβαια αντικριστώ του κυρίο έχουν ε, πρόεδρος και θέλω να σας πω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, ε, αν ε, θέλετε να σεβαστούμε το χρόνο, κάπως θα πρέπει να περικόψουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν θα προβώ σε συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε άλλη μισή ώρα για τους ε, υπόλοιπους τρεις προσκεκλημένους για να μην έχουμε συζήτηση στο δεύτερο πάνελ. Ξέρω ότι όταν ένας εμπειρογνώμονας ε, πιέζεται για να εκφράσει τις ιδέες του μέσα σε 10 λεπτά, φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά προσπάθησα να περιγράψω μια προσέγγιση σε περισσότερε συνεργασία σήμερα. Όλα όσα λέγονται σήμερα διαβιβάζονται στις αρμόδιες στην Ομαδία Εργασία για την ασφαλεία στην κοινωνική χώρο και ε, στους εισηγητές της κυρίας Επιτροπής, της Καθήλια Αρμόδια Επιτροπής και στις υπόλοιπες επιτροπές. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο για συζήτηση, μη φοβάστε γιατί ο χρόνος που επενδύουμε χρησιμοποιείται ορθά. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο πάνελ. Ελπίζω να συμφωνείτε. Λοιπόν, η προστασία των δεδομένων είναι ένα από τα κύρια θέματα που ασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστηρίζουμε το λειτουργήμά σα. Εμεί ε, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Χάνστιξ ε, θα αναφερθεί στο θέμα τη προστασίας ε, των δεδομένων των πολιτών. Θα σα δώσω το λόγο για να αναφερθείτε στι νομικέ πτυχέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω αυτή την ακρόαση για τις κυβερνοπιθέσεις συναντήσεις των πληροφοριών και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια δικαίου για πολύ καιρό. Ο όρος κυβερνοχώρος αναφερόταν σε μια πολύ μακρινή πραγματικότητα και ίσως εφευρέθηκε για να υπονοεί ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο χώρο. Αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι δεν είναι τόσο μακριά πλέον ο χώρος αυτός. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο γενικά και οι κυβερνοεπιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο. Αλλά θεμελιώδε νομικές αρχές θα πρέπει επίση να ισχύουν και στον κυβερνοχώρο, όπως ισχύουν στον πραγματικό κόσμο και εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Αυτό ισχύει και για την έννοια του εγκλήματος, αλλά και για την καταπολέμηση και την ε, πρόληψη του εγκλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν ε, υπάρχει καθολικό μέσο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να καλύπτει όλες τις πτυχές καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος. Η απόφαση του Συμβουλίου 2005-222 καλύπτει μόνο την προσέγγιση των ορισμών ορισμένων αδικημάτων στον κυβερνοχώρο και δεν ε, καλύπτει όλο τον αριθμό των αδικημάτων, ε, ούτε βρίσκεται τους τρόπους για την καταπολέμηση των κλίματων στον κυβερνοχώρο ε, ούτε θέτει τι δικλείε ασφαλεία που χρειάζονται. Οι σημερινοί κανόνε για την προστασία των δεδομένων για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη αποτελούν σήμερα ένα patchwork ειδικών κανόνων και ένα γενικό πλαίσιο στον τομέα αυτό είναι περιορισμένο παιδί εφαρμογή καθώς ε, εφαρμόζεται μόνο στις ροές δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ε, μετά την Λισαβόνα έχουμε μια μεγάλη, μεγάλη για την προστασία των δεδομένων ε, λόγω της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της συνθήκης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επίσης εξηγεί τη δουλειά που έγινε για την αναθεώρηση της σημερινής ε, οδηγίας προστασίας των δεδομένων. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει μια συνολική προσέγγιση, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και όλων των τομέων ε, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του προηγούμενου τρίτου πυλώνα. Αστυνομία και δικαιοσύνη, αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε περισσότερη αποτελεσματικότητα και το έχω πει και στο παρελθόν. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν είναι ο καιρός τώρα να επανεφεύρουμε την προστασία των δεδομένων. Έχει εφευρεθεί και τώρα να γνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αντίθετα, πρέπει να δοθεί καλύτερη προσοχή στο να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική στην πράξη την προστασία των δεδομένων και αυτό σημαίνει να στήσουμε περισσότερο στην εφαρμογή των αρχών της ε, προστασίας των δεδομένων και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων για τους οποίους αφορούν τα δεδομένα. Επίσης, ε, η συμπερίληψη των αρχών privacy by design και της λογοδοσίας είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό γιατί θα συνεισφέρει σε ένα πιο βιώσιμο κυβερνοχώρο. Πολλά παραδείγματα, σήμερα το απόγευμα μας έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωση αλλά επίση είδαμε ότι μακροπρόθεσμα προγράμματα όπω το ψηφικό θεματολόγιο και το πρόγραμμα τη Στοκχόλμης τόνισαν τη σημασία τη καταπολέμηση του κυβερνού εγκλήματο και η προτινόμενη οδηγία που συζητείται τώρα αποτελεί ένα βήμα προ τα μπρο. Δεν είναι μεγάλο βήμα, αλλά είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Και είναι σαφές το επεξηγηματικό μνημόνιο ότι η πολιτική επιλογή που επιλέχθη ε, θα στοχεύει στην, στοχεύει στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης απόφασης πλαίσιο. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και θεματικά. Παρ' όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα να αναφέρω παρόλα αυτά την εφιστάμενη κοινωτική νομοθεσία η οποία ισχύει για να διασφαλίσει ότι δεν έχουμε ούτε την αγρία δύση στον κυβερνοχώλο, αλλά ούτε και ένα χώρο μεγάλο δελφού. Αν ε, δούμε τη χαρτί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το μήνυμα είναι ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα ε, σεβασμού τη ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή ε, και τη επικοινωνία. Το καθένα έχει δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν τέτοια δεδομένα πρέπει να τη χάνουν δίκαιες επεξεργασίες για συγκεκριμένους σκοπούς και βάσει της ε, συνένεσης των διαφορεμένων ατόμου ή βάσει κάποιες άλλες νόμιμης βάσεις, δυνάμει της νομοθεσίας. Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ε, και τον αφορούν και έχει δικαίωμα διόρθωσης. Συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες θα υπόκειται σε έλεγχο από μια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό ισχύει και στον κλειμένο χώρο και στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον χώρο. Η επίσης η σημερινή οδηγία προστασία των δεδομένων και οι υπόλοιποι κανόνες οι σχετικοί έχουν ισχυρό ρόλο για την πρόληψη του εγκλήματος στον κυβερνό χώρο καθώς ε, οι ελεγκτές ε, υποχρεώνονται να αναλύουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να προωθήσουμε. Τώρα, αν δούμε την ασφάλεια δικαίου ευρύτερα, υπάρχει μια γκάμα νομοθετημάτων που κατά κάποιο τρόπο συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον χώρο. Σύμβαση της Βουδαπέστης, η οποία ακυρώθηκε από τα 15 από τα 27 κρατημέλη, όπως γνωρίζω, δεν ε, είναι πάρα πολύ καλό βέβαια το σκορευτό, το σκορευτό έχουμε επίσης διατάξεις ε, σχετικά με την ε, εμπιστευτικότητα ε, όπου εκεί αναφέρονται κάποια θέματα σχέση με τις παραβιάσεις των δεδομένων, το απόρριτο κτλ. Η οδηγία για την διατήρηση των δεδομένων έχει δεκτεί ε, μεγάλη κριτική. Επίσης υπάρχουν ε, υφιστάμενες νομοθεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη και έχουμε και μέσα συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας βάσει ε, των κεφαλαίων 4 και 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένα μπορούν να εφαρμοστούν και για το εγκλήμα στον κεφαλαίο χώρο. Και υπάρχει και μια γκάμα δραστηριοτήτων σε ευρύτερο πεδίο σχέδιο δράση για την προστασία τη ε, υποδομή ζωτική σημασία, συνεργασία μεταξύ των ΣΕΡΤΣ, ε, η ΕΝΗΣ αναφέρθηκε, η Europol και η Eurojust ε, και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Κρατών Μελών έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην ανθεκτικότητα ασφαλείας των υποδομών και επίσης ε, ε, η Ευρωπαϊκή ΔΙΤ για την ανθεκτικότητα. Τώρα, μιλούμε για ασφάλεια δικαίου. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο των πολλαπλών νομοθετημάτων που εφαρμόζονται ε, οι αρμόδιοι Επίτροποι για την Προστασία των Δεδομένων και η Ομάδα Εργασία Αστυνομική Συνεργασία και Δικαιοσύνη έχουν δώσει κάποιε ενδείξει που μπορεί να είναι χρήσιμες, δηλαδή ε, να Έχουμε πρόληψη του ορισμού των αδικημάτων ε, που καλύπτονται από τα εκτελεστικά μέτρα της σύμβασης από το να ε, μην είναι υπερβολικά ευρεία σε σχέση με το τι τίθεται στην ίδια τη σύμβαση επίσης. θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ορισμό των κατηγοριών που συλλέγονται και ενταλλάσσονται στην δική νομοθεσία είναι ανάλογη και επίση να μην υπάρχει επικάλυψη στα κράτη-μέλη σε σχέση με τι διατάξει για το πάγωμα των δεδομένων που έχουμε στη σύμβαση. Και σε σχέση με τη διατήρηση των δεδομένων υπό την οδηγία 2006-24. Τελικά σχόλια. Το να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση των κλίματων στον κυβερνοχώρο δεν απαιτεί συνεχή και συστηματική εποπτεία των χρηστών στο ίντερνετ. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου τέτοια εποπτεία αφήνεται στους ΕΣΠΗ και άλλους ε, παρόχους ε, στη βάση ε, του πεφωτισμένου αυτοσυμφέροντος η συστηματική γνηλάτιση των χρηστών αποτελεί πραγματική παραβίαση των θεμελιωδονομικών ε, αρχών και δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μόνο να έχουμε στοχευμένα μέτρα όπου απαιτούνται και να είναι αναλογικά με όλες τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό ισχύει και στον τομέα του κλίματος του κυβερνοχώρου. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Πίτερ Χάστινγκς, ευχαριστώ για την θαυμάσια επισκόπηση ε, και τώρα χαίρομαι πολύ διότι έχουμε σήμερα εδώ την κυρία Μαρία Καϊάφα, καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης η οποία είναι σαφώς μία από τις ε, πιο γνωστές ε, καθηγήτριες στον τομέα της πρωτοβουλίας ποινική πολιτικής στην Ευρώπη και ε, της δίνω τώρα το λόγο. Την ευχαριστώ που ε, σήμερα μπόρεσε να έρθει στην ε, συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ κυρία Χολμάγερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ε, ευγενή πρόταση να έρθω εδώ σήμερα διότι ε, θα ασχοληθώ με ε, την ε, πρόταση της οδηγίας και ιδίως ε, ποια πρέπει να είναι η βάση των επιλογών που θα γίνουν στα πλαίσια των βασικών αρχών του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το θέμα αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με ε, την ε, έντολη ότι ε, η ποινική νομοθεσία θα πρέπει να σέβεται τις, τα υψηλά επίπεδα δημοκρατικής νομιμοποιήσεως, το κράτος δικαίου και να βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας ελευθερίας και των βασικών νομικών αρχών. Γι' αυτό και θα ασχοληθώ με ε, την ε, παράνομη ε, παρέμβαση σε στοιχεία ηλεκτρονικά στο άρθρο 6 και την παραγωγή πώληση εργαλείων που χρησιμοποιούνται για παράνομες επιθέσεις στα κομπιούτερ κομπιούτερ καθώς και σε ένα γενικότερο πλαίσιο διότι η πρόταση ε, αλλάζει ε, τη διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υποκίνηση, την ε, βοήθεια, την προσπάθεια και ιδίως με τις εφαρμόσιμες πυρώσει. Ξεκινώντας λοιπόν με το είδη συμπεριφορών που προβλέπονται εις την απόφαση πλαίσιο, πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόταση οι οδηγίες διευρύνει ε, ε, ε, την, αρχή της παράνομης προσβάσεως σε συστήματα πληροφοριών και παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας. Αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορέσουν να εφαρμόσουν ορισμένους περιορισμούς βάσει της αρχής ultima ratio. Διότι αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τα συστήματα πληροφοριών από την ε, άκρατη ποινικοποίηση. Και γι' αυτό μπορούμε απλώς να ε, χαιρετήσουμε την πρόταση αυτή του Συμβουλίου η οποία επαναφέρει ε, την παραβίαση των μέτρων ασφαλείας σαν προϋπόθεση για να βεβαιωθεί η παράνομη πρόταση πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά οι ε, διατάξεις που αναφέρονται στα παράνομα συστήματα και στην ε, παράνομη παρέμβαση ε, στα στοιχεία δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με την αρχική απόφαση πλαίσιο και γι' αυτό δεν θα τα σχολιάσω αλλά βλέπω ότι όσον αφορά την νέα διάταξη που αναφέρεται στην παράνομη ε, επέμβαση των, ε, σε στοιχεία που δεν μεταδίδονται δημόσια με τεχνικά μέσα. Το ε, Συμβούλιο της ε, Ευρώπης και η σχετική σύμβαση επιτρέπει στα κράτη να ποινικοποιήσουν τη συμπεριφορά η οποία οφείλεται σε ε, παράνομη πρόθεση. Ε, αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει τα, τις ίδιες προϋποθέσεις και γι' αυτό υπάρχει μία σαφής διάταξη που επιτρέπει πρέπει να εφαρμοστεί νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο και η σύμβαση σχετικά με το κυβερνοέγγραμμα επαρκεί ε, για να αποδειχθεί η ανάγκη για έναν πιο εκτενή ορισμό ε, της παρεμβάσεως, interception. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να πρινικοποιήσουν την παραγωγή, πώληση και ε, ιδιοκτησία οποιοδήποτε μέσου το οποίο συμπεριλαμβάνει και λογισμικό που μπορεί να προσαρμοστεί ή έχει προβλεφθεί ε, για να εφαρμόσει αυτά ε, τα αδικήματα. Στα άρθρα τη συνθήκης βλέπουμε ότι υπάρχει μια σωστή επιλογή από το Συμβούλιο της Ευρώπης που περιορίζει την ποινικοποίηση στην ε, διανομή των ε, δυνητικά επικινδύνων ε, μέσων ενώ μία από τις συνθήκες Συμβουλίου της Ευρώπης και οι σχετικοί περιορισμοί δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρώπη γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να συνάδει ε, το, η, ρύθμιση του Συμβουλίου της Ευρώπης με ε, την προτινόμενη οδηγία. Ε, θα υπάρχει προσπάθεια να ποινικοποιήσουμε και την σύνδρομη και δεύτερον τα κράτη-μέλη πρέπει να ποινικοποιήσουν Παρακαλούμε την ομιλήτρια λίγο να επιβραδύνει την ε, ανάγνωσή της. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη πρέπει να ποινικοποιήσουν τις προσπάθειες ε, χωρίς εξαιρέσεις ε, ε, σύμφωνα με ε, την σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα ενώ από την άλλη πλευρά εξαιρείται ε, από το αδίκημα το άρθρο 7 και ε, υπάρχει επίσης περιορισμός των προσπαθειών σύμφωνα με την πρόσφατη ε, πρόταση του Συμβουλίου όσον αφορά τα αδικήματα των παρανόμων ε, παρεμβάσεων στα συστήματα και στα στοιχεία αλλά βλέπουμε ότι ε, έχουμε πολύ βασικές διαφορές στο επίπεδο του άρθρου 2D όσον αφορά την ε, καταστολή της εγκληματικότητας όπου τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε παραβίαση τιμωρείται με ε, φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών εκτός από την αρχή της αναλογικότητας αυτό, αυτή η ποινή αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άκαμπτη ε, και δεν ε, ακολουθεί την ιδέα μεγαλύτερης ευελιξίας. Παραδείγματος χάρη ένα το επίπεδο φυλάκισης από ένα έως τρία έτη. Είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε την αναλογικότητα του, της αποφάσεως πλαίσιο ε, κατά τρόπον ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν και να σταθμίσουν την σοβαρότητα της αξιόπινης πλάξεως και ε, να μην υπάρχουν πιο αυστηρές ε, κυρώσεις που θα περιορίσουν τη δυνατότητα διεκριτικής ευκαιρίας των κρατών μελών ή στον καθορισμένο τους. Επίσης η στον καθορισμέ τους επισης η διαταξη του άρθρου 10 ε, διευρύνει την απαρίθμηση των ε, επιβαρυντικών συνθήκων και μπορεί να οδηγήσει ε, σε μία ποινή τουλάχιστον των 5 ετών αντί για δύο 5 σύμφωνα με το άρθρο 7. Ε, και γι' αυτό η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ζήτησε από τους Υπουργούς να ζητήσουν καθοδήγηση για να αποφύγουν ένα διέξοδο μέσω των ε, ε, εξηγηματικών πράξεων και δεύτερον μέσω μίας αναδιαμορφώσεως των επιβαρυντικών συνθήκων ε, και ε, της, ε, του περιορισμού των κυρώσεων σε αδικήματα που αναφέρονται εις την παράνομη επέμβαση στα συστήματα και στοιχεία. Βλέπουμε εδώ ότι το προήμιο της οδηγίας ε, αναφέρεται στους βασικούς λόγους που οδήγησαν στις επιλογές που έγιναν για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία και να μπορέσει ε, να ε, υπάρξει μία διατύπωση ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στις πράξεις αυτές αντί να επεκταθεί το ισχύον ποινικό δίκαιο σε αυτές τις περιπτώσεις στην, ε, ε, άλλωστε η πρόταση για μία οδηγία εξασφαλίζει προστασία ε, των βασικών δικαιωμάτων και εδώ δεν ε, υπάρχει συμμόρφωση στην ανάγκη του Lex Certa που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση και θα πρέπει να υπάρξει και ο σαφής χαρακτήρας των ε, επουσιωδών περιπτώσεων οι οποίες δεν ποινικοποιούνται. Η αρχή της αναλογικότητας επίσης υποθάλπιται γιατί η αναλογικότητα δεν εξυπηρετείται όταν τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό των εφαρμοστέων κυρώσεων. Τέλος, θα πρέπει να ανησυχούμε για ε, μία ποινικοποίηση των προκαταρκτικών ε, πράξεων όπως η παραγωγή εργαλείων που ε, θα χρησιμοποιηθούν για τη δυνητική επέμβαση και την εκτέλεση των αξιοπίνων πράξεων διότι είναι προφανές ότι η ποινικοποίηση όλων αυτών των συμπεριφορών μπορεί να βασιστεί σε υποκειμενικά κριτήρια και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει τη δυνατότητα να περιοριστεί ο τομέας αυτός και συνδυάζεται με ε, την αναγνώριση της ε, εξοεδαφικής ε, δικαιοδοσίας δημιουργεί μία δυσχερή κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή ultima ratio και τις αρχές της νομιμότητος, της αναλογικότητος και του σεβασμού της συνεκτικότητας σε κάθε κράτος μέλος. Δηλαδή θα πρέπει να ε, ε, υπάρξει ορισμός των παρανόμων επεμβάσεων, των τεχνικών μέτρων, των ε, επουσιοδών περιπτώσεων, των επιβαρυντικών συνθήκων, καθώς επίσης και διεύρυνση του άρθρου 7 που αναφέρεται στις προκαταρκτικές ενέργειες αν δεν καταργηθεί αυτή η διάταξη. Εις ε, το παράτημα της παρουσιάσεώς μου θα βρείτε έναν κατάλογο συγκεκριμένων προτάσεων διότι θεωρώ ότι αυτές οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μόνο έτσι θα εξυπηρετηθούν οι βασικές αρχές του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιτευχθεί ο στόχος δηλαδή να τοποθετηθεί το άτομο εις το επίκεντρο των ε, ε, δραστηριοτήτων. Οι λαοί της Ευρώπης προσβλέπουν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σημειώσει αυτές τις ενέργειες. Κυρία ε, Καϊάφα, προσπαθήσατε πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια να μας παρουσιάσετε το κείμενό σας. Εγώ σας ευχαριστώ σαν εισηγήτρια και θα επανέλθω για διάφορα θέματα τα οποία αναφέρατε στην έκθεσή σας και τα οποία θα μπορέσω να συζητήσω και με τους άλλους και εισηγητές για να επανέλθω. Λοιπόν, ε, και τώρα ερχόμαστε προς το τέλος. Ε, ζητήσαμε από τους διερμηνείς να παραμείνουν ακόμη 10 λεπτά. Τους ευχαριστώ γιατί σήμερα ε, κάνουν εξαιρετικές προσπάθειες να παρακολουθήσουν την ταχύτητα των ομιλητών, πράγμα το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση, γι' αυτό και τους ευχαριστώ λέγει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ επίσης που θα μείνουν ε, λίγο ακόμη μαζί μας. Και ε, τώρα θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Τζο Μακνάμι της Ευρωπαϊκής Ομάδας Προστασίας Ψηφιακών Δικαιωμάτων που είναι μία ομάδα ε, που προασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών ή στην κοινωνία μία της πληροφόρησης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας δίνω το λόγο. Θα προσπαθήσω να κάνω την παρουσίασή μου στο δυνατόν γρηγορότερα χωρίς και να τρελάνω τους διερμηνείς. Θα παραλείψω την εισαγωγή γιατί έχουν υποθεί πολλά από αυτά που ήθελα να πω Θα ήθελα να σας πω ότι είναι αυτό το θέμα από τα σπουδαιότερα που, ε, με τα οποία έχω ποτέ ασχοληθεί και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα θέμα θέλω να θίξω, αυτό που ανέφερε και η κυρία Χολμάγερ σε προηγούμενες στιγμές Η θέση της Ένωσης για τις επιθέσεις έναντι, εναντίον μάλλον ηλεκτρονικών συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και θα σας το αποδείξω τώρα. Οι επιθέσεις κατά ηλεκτρονικών συστημάτων είναι κάτι γνωστό. Έχει γίνει η επίθεση κατά του Ιράν, το Stuxnet, και εδώ γίνεται και ένας πόλεμος διευθύνσεων και domain names που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την καταστολή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ένωση. Μέχρι πρόσφατα δεν χρησιμοποιήθηκε η νομολογία που υπάρχει κατά εταιριών και υποδομών που υπάρχουν στο ίντερνετ. Υπάρχει ο νόμος Protect IP και COICER. Στις Ηνωμένε Πολιτείες δίνεται καμιά φορά το δικαίωμα σε εταιρείε να ε, χρησιμοποιήσουν δεδομένα από συστήματα που είναι εκτός της δικαιοδοσίας τους. Και επομένως παραμένει το θέμα του κατά πόσον είναι βιώσιμοι οι ορισμοί που δίνει η οδηγία αυτή. Λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιτρέψει την επίθεση κατά ηλεκτρονικά. Επομένως πρέπει να δούμε σαφέστερα τι είναι εγκληματική πράξη. Πέρυσι το domain name moon.com απαγορεύτηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθουσαν λέει να καταπολεμήσουν έτσι δεκάδες ιστοσελίδων παιδοπορνογραφίας αλλά έτσι κατήργησαν και αθώες ιστοσελίδες κατηγορώντας 84.000 χρήστες για εγκλήματα κατά της αθωότητος των παιδιών. Πέρυσι επίσης υπόθηκε ότι από τη Unilever ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος μέσω της κατάργησης domain names. Το Συμβούλιο πριν από τρεις εβδομάδες δέχτηκε αυτή την προσέγγιση και κάλεσε τις χώρες μέλη να προασπίσουν την ακαιρεότητα του ίντερνετ. Ο Ισπανός εισηγητής ξέρει τι σημαίνουν όλα αυτά από την εμπειρία του. Ένας Βρετανός πολίτης που ζούσε στην Ισπανία είχε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που ειδικευόταν σε ταξίδια στην Κούβα και από μια μέρα στην άλλη εξαφανίστηκαν οι ιστοσελίδες του. Δεν είχε δραστηριότητα στις Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε συμφέροντα στις Ηνωμένε Πολιτείε και όμως είχε μπει σε μαύρο κατάλογο από το Υπουργείο Οικονομικών των ΙΠΑ και η εταιρεία που του είχε χορηγήσει την πρόσβαση την αφαίρεσε και έμεινε χωρίς καθόλου έσοδα. Πιο πρόσφατα οι Ηνωμένε Πολιτείε κατήργησαν και άλλο όνομα ισπανικής εταιρείας με την κατηγορία ότι παραβίαζε πνευματικά δικαιώματα κατηγορία που την απέρριψαν ήδη τα ισπανικά δικαστήρια. Εν τω μεταξύ οι θεώρησαν ότι οτιδήποτε καταλήγει σε τελεία ακόμη είναι αμερικανικής δικαιοδοσίας. Επομένως τα προβλήματα που αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πραγματικά. Υπονομεύεται όντως το ίντερνετ Τι κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα. Όχι ό,τι θα νόμιζε κανείς. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν έχουν διαμαρτυρηθεί, αλλά έχουν ενθουσιωδώς δεχτεί αυτές τις επιθέσεις. Και η αμερικανική πρόταση μιας κοινή ενωσιοαμερικανικής κατάργησης ονομάτων αν γίνει δεκτή θα σήμαινε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να παρέμβουν σχεδόν οπουδήποτε σε όλο το χώρο που καλύπτει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ονομάτων. Η ανακοίνωση της Κομισιόν απορρίφθηκε από την Σουηδική Προεδρία αλλά επανυποβλήθηκε υπό την Ισπανική Προεδρία και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών και το Υπουργείο Γενικών Υποθέσεων το 9. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στους προμηθευτές πρόσβασης και λέει ότι εκτός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοια δικαιώματα κατάργησης ονομάτων γιατί συνιστούν έγκλημα. Άρα εδώ η κατάσταση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα δίνει στον εαυτό της τη δικαιοδοσία παράνομα να κατακρατά και να απαγορεύει ονόματα και προτείνει κυρώσεις για την παράνομη κατάργηση ονομάτων. Το cloud computing θέτει ένα πρόβλημα περιεχομένου του ίντερνετ και πρέπει το κοινοβούλιο να το δει και αυτό. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το περιεχόμενο του ίντερνετ πέρυσι είχε δίκιο. Αλλά αν οι Ευρωπαίοι χρήστες βγαίνουν στο ίντερνετ χωρίς καμία νομική βεβαιότητα και μόνο να μαντέψουν μπορούν τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχει ο προμηθευτής της πρόσβασής τους ή ποια είναι η πολιτική της εταιρείας που τους δίνει τις υπηρεσίες αυτές, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Η οδηγία δεν είναι πολύ λανθασμένη, αλλά γιατί όντως πρέπει να προστατευτεί η πληροφόρηση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εκείνοι δεν κάνουν το σωστό, αλλά εμείς το κάνουμε, αφού κάνουμε το ίδιο πράγμα. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς και αυτούς που κάθονται εδώ αλλά και ε, τους ακροατές που άντεξαν μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την κατάρτιση μίας ε, λογικής οδηγίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε όλοι οι ομιλητές τα κείμενά σας γραπτά. Ορισμένοι εξ τα είχαν ήδη για να μπορέσουμε να μελετήσουμε ακριβώς αυτά τα οποία μας ε, είπατε και θα σας παρακαλούσα να ε, παραμείνετε ακόμη για ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες έχει ε, και η συγγήτρια και ο σκιώδης εισηγητής και γι' αυτό σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έμειναν μέχρι το τέλος ε, και ε, εμπλούτησαν το, τη συζήτηση. Ευχαριστώ τους διερμηνές που έμειναν ως τώρα και ε, όντως πρέπει να σας χειροκροτήσουμε γιατί κάνατε εξαιρετική δουλειά. Καλό βράδυ.